I, normally I don't use it, but sorry, please. Oh, eh, sorry, please. Μπορούμε να αρχίσουμε τώρα, αλλά να καθίσετε παρακαλώ. Λάβετε θέσεις. Μπορούμε να αρχίσουμε αν δεν απατώμε. Ήρθατε όλοι και όλες, εντάξει. Λοιπόν, θα αρχίσουμε αν δεν απαντώμε με το πρώτο σημείο. Πάμε λοιπόν, έγκριση της ημέρησης διάταξης, πρώτο σημείο στην ημέρησια διάταξη. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, εγκρίνουμε το πρώτο σημείο. Πάμε στο δεύτερο σημείο, έχετε παρατηρήσει τα πρακτικά της συνεδριάσεως της 12ης Νοεμβρίου. Αν δεν έχετε, συνεχίζουμε. Τρίτο σημείο, ανακοινώσει της Προέδρου. Πρώτα απ' όλα έχουμε διαρμηνία για Ιταλικά, Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Τσεχικά, Πολωνικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Ουγγρικά και Στονικά. Και έχουμε web streaming όπως πάντα, μεταδιδόμαστε μέσω διαδικτύου. Οι αποφάσεις των συντονιστών της 12 η Νοεμβρίου έχουν αποσταλεί όλα τα μέλη της Επιτροπής μέσω email τις επόμενες μέρες. Εγκρίθηκαν επίσημα διότι δεν είχαμε αντιρρήσει μέχρι τις 18 Νοεμβρίου που είχε διοριστεί σαν προθεσμία. Θα ήθελα να καλωσορίσω την, την, την το νέο μέλος της Επιτροπής μας. Καλώς ήρθατε. Η κυρία Τερέζα. Τερέζα Χεμένε Μπαρμπάτ από την ΑΛΤΕ που αντικαθιστά την κυρία Μάουρα Μπαρανταριάν. Χαιρόμαστε πολύ για την παρουσία σας εδώ και ευχόμαστε καλή δουλειά, καλή συνεργασία. Ε, κάποια πράγματα να σας πω, εν συντομία. Βλέπω υπάρχει κάποια ταραχή στην αίθουσα. Το πρώτο που έχω να πω στο Στασβούργο με κάποιους συναδέλφους που είναι παρόντες, όχι πολλούς, είχαμε ενδιαφέρουσα συνάντηση με την ε, αντιπροσωπεία του Μασρέκ όσον αφορά τα θέματα της πολιτισμικής κληρονομιάς. Εγώ συμπρόεδρευσα μαζί με τον συνάδελφο Ανδρέα Κοτσολίνο, αντιπρόεδρο ε, της Επιτροπής για το Μασρέκ. Έγινε μια ενδιαφέρουσα ακρόαση όσον αφορά τα θέματα τα πολύ δύσκολα και θα έλεγα την καταστροφική κατάσταση όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά που καταστράφηκε στη Συρία. Κάναμε μια ακρόαση, ακούσαμε την δόκτωρ Αλή Τσεκμούς τη υπηρεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων στη Συρία, είναι αρχαιολόγο από τη Συρία ε, που είναι ε, σε εξορία στη Γαλλία. Ε, πολύ σημαντική προσωπικότητα και έκανε κάποιες προτάσεις που υπογραμμίζονται σε ένα έγγραφο που δείχνει το έγγραφο την κοινή θέση δύο διαφορετικών ενώσεων και όπου εκεί, εκεί συμμετέχουν ε, Σύρια αρχαιολόγοι. Ήρθαμε σε επαφή μαζί τους, ε, ε, είδαμε κάποιες διαφάνειες πώς ήταν η κατάσταση στις αρχαιότητες και πώς είναι τώρα. Είδαμε περίπου 12 τοποθεσίες, 12 αρχαιολικούς τόπους που είτε καταστράφηκαν ή υπέστησαν μερική καταστροφή ε, προτάθηκε σε εμά την ε, αντιπροσωπεία του Μασρέκ και θα θέλαμε να συνεργαστούμε μαζί τους περαιτέρω για το τι θα κάνουμε, ζητούσε ένα είδος μονάδα κρίσεων, crisis units, που να συμμετέχουν εμπειρογνώμονες και Συρίοι και Ευρωπαίοι για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε, να εξετάζουμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, ποια παρέμβαση θα μπορούσε να ε, λάβει η χώρα, ποια είναι η τεχνογνωσία για τα θέματα και τι να κάνουμε από τη στιγμή που όπως ελπίζουμε και ευχόμεθα να λήξει η σύγκρουση κατά κάποιο τρόπο και να προετοιμάσουμε τη μετέπειτα κατάσταση. Εγώ υπογράμμισα αυτά που κάναμε στην Επιτροπή Πολιτισμού, ότι είμαστε διαθέσιμοι, είπα πόσο δραστηριοποιούμεθα στον τομέα και ουσιαστικά στο τέλος αποφασίστηκε να γίνει μία εξέταση των δυνατοτήτων που ανοίγονται μπροστά μα, ζητώντα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κάποια ε, κινητοποίηση και μετά σε ενημερώσουμε. Όμω νομίζω ότι περισσότερη συνεργασία μαζί με τι διάφορε αντιπροσωπείε και αυτή και του Μαγκρέμπ, διότι μιλάμε και για τι ε, προοπτικέ περισσότερων σχέσεων με τις χώρες της Μεσογείου και της περιοχής των Βαλκανίων και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Άλλη ενημέρωση που έχω να σα κάνω. Τα πρακτικά η ε, έκθεση για την αποστολή μας στη Φλωρεντία σας έχει μοιραστεί πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Να επισημάνω ότι από πλευρά του Ινστιτούτου του, του Φιδέντς της Φλωρεντίας που είναι ένας, ένας φορέας ύψης της ποιότητας αριστείας. Εκεί στο Ινστιτούτο γίνεται εξέταση της περιπτώσεως με την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου να δημιουργηθεί ένας νέος τομέας, μία ανωτάτη σχολή μελετών για την υπερεθνική διακυβέρνηση. Τα μεγάλα θέματα αφορούν αυτή την υπερεθνική διακυβέρνηση και είναι ενδιαφέρον τομέας έρευνα. Θα ήθελα να σας πω εν συντομία και κάτι άλλο, ότι ήταν σημαντική συνεδρίαση και η επαφή που είχαμε στις 3 ε, Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους που συμμετείχαν, 23 συνάδελφοι συμμετείχαν ε, πλήρη με 16 πλήρη και οι ε, υπόλοιποι ήταν πραγματικά μπορεί να κάνετε λίγη ησυχία παρακαλώ λίγη ησυχία και μετά ήρθαν 18 εθνικοί βουλευτές και εκπρόσωποι εδώ των Βρυξελών των Εθνικών Κοινοβουλίων εκπροσωπώντας 12 χώρες πρέπει να πω ότι ήταν μια συνάντηση, μια διάσκεψη η οποία έδωσε, μας έδωσε μεγάλη ικανοποίηση και σε εμά και σε εσά για κάποιου λόγου. Πρώτα απ' όλα, διότι ήταν μια διάσκεψη που κατέδειξε τη βούληση που έχει η Επιτροπή μα και το Κοινοβούλιο βέβαια, σύμφωνα με, με τον τρόπο που πρέπει να ακολουθείτε, να συζητούμε άμεσα με τα εθνικά κοινοβούλια και να ενισχύσουμε στα εθνικά και ευρωπαϊκά θεματολόγια τα ζητήματα του πολιτισμού και της παιδείας και των πολιτικών για τους νέους και ακολουθούμε ε, ανιούσα και κατιούσα πορεία στον αφορά τι ε, επαφέ που ακολουθούμε στα διάφορα επίπεδα. Πρώτη φορά συναντήθηκαν κάποιοι βουλευτέ μα με συναδέλφου από άλλε χώρε, άρα ισχύσαμε κάποιε σχέσει και πρέπει να σα πω ότι το Youth Forum, το European Youth Forum, ε, δέχτηκε τι ευχαριστίε μα διότι πήρε πολύ σοβαρά τον διαθρωμένο διάλογο και έχουμε συναδέλφους που πήραν το λόγο και σφαίρ όλους εκείνους ε, που πήραν το λόγο τους ευχαριστώ που μίλησαν για τις σχέσεις που πρέπει να έχουμε με τους νέους και για τις προπτικές για το 2020 και ήταν χρήσιμο να ακούσουμε ε, ποια ήταν τα θέματα που θεωρούν πάρα πολύ σημαντικά σήμερα. Η Προεδρία του Λουξεμβούργου πέραν του ότι υπενθύμησε ότι ενεκρίθη στο τελευταίο Συμβούλιο μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Συμβουλίου ετοίμασε έκθεση όχι μόνο για τους νέους και τη σχέση με τους νέους, αλλά για μεγαλύτερη προσοχή που θα πρέπει να δοθεί στη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή, διότι αυτή η ριζοσπαστικοποίηση και αυτή η αποξένωση ε, είναι κάτι κακό. Είδαμε και σε εκλογέ δεν συμμετείχαν πολλοί και η ριζοσπαστικοποίηση των νέων είναι ένα πρόβλημα. Δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει μια αύξηση τη αποστασιοποίηση. Αυτό είναι ένα θέμα που ε, το τόνισαν όλοι και ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να βρουν απο... απαντήσεις πιο σημαντικές, να επενδύσουν περισσότερο στα προγράμματα αυτά που εδράζονται από αυτών των θεμάτων. Εμείς εργαζόμαστε σαν Επιτροπή Πολιτισμού, αλλά πρέπει να δοθεί μια απάντηση εν γέννη. Μια άλλη πτυχή που διεφάνει ήταν ότι χρειάζεται περισσότερη επένδυση, αν θέλετε μεγαλύτερη προσπάθεια και πόρη για την, την ένταξη, για την παιδεία, και κυρίως οι μετανάστες να ενταχθούν και το Συμβούλιο Υπουργών στο Συμβούλιο Υπουργών του Λουξεμβούργου είπε ότι έγινε μια πρόταση ούτω ώστε να είναι εκτός του Συμφώνου Σταθερότητας τουλάχιστον οι ποσοστώσεις που αφορούν αυτό διότι μία από τις στοιχείες ασφαλείας διότι Λοιπόν, το θέμα της ασφαλείας θα πρέπει να καλυφθεί. Αυτή η πρόταση ε, υποστηρίχθηκε από κάποιες χώρες, από την Ιταλία και το τονίζω γιατί ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Βάλαμε στο επίκεντρο το διαπολιτισμικό διάλογο και αυτό εξετιμήθη. Η παιδεία που εντάσσει όλους, περιλαμβάνει όλου. Πολλοί θεώρησαν ότι η οικονομική κρίση και οι δυσκολίες όχι μόνο οδηγούν σε ανεργία των νέων που είναι υψηλή, αλλά μας οδηγεί και σε ολιστική προσέγγιση που απαιτείται. Ανάκτηση των διαφόρων ε, ε, ε, των δεξιοτήτων και συμμετοχή στην εθελοντική εργασία και στον αθλητισμό. Να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην εγγύηση αφορά τους νέους για τις δεξιότητες και για την απασχόληση. Άρα και πιο, απαιτείται πιο εγκάρσια προσέγγιση. Κάτι άλλο σημαντικό. Και οι νέοι ζήτησαν να αναγνωριστεί καλύτερα ο διαθρωμένος διάλογος για τα δικαιώματά τους, για την άμεση συμμετοχή τους, για την δυνατότητα του συνεταιρίζεστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Μόνο τρία συμβούλια των νέων συμπεριελήφθησαν στα κράτη-μέλη για την προετοιμασία των εγγυήσεων για τους νέους. Λοιπόν, αυτή ήταν μια μεγάλη συζήτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είδαμε ότι υπάρχει μεγάλη δέσμευση και αφοσίωση για συγκεκριμένους στόχους, για ότι ενθερμίζεται τις ανησυχίες προτεραιότητες. Θέλαμε να έχουμε κάτι παραπάνω, πιο στέρεο, πιο συγκεκριμένο. Το μόνο που θεωρώ ότι είναι σημαντικό να επενθυμίσουμε, ένα από τα πράγματα τα πιο σημαντικά που πρέπει να επενθυμίσουμε από πλευράς της Επιτροπής είναι ότι θεωρώ ότι ότι κάτι επεξεργάζονται, δεν ήταν σαφέ, επεξεργάζονται κάτι. Προγράμματα ίσως που θα μπορούσαν μαζί με τα πανεπιστήμια και τα σχολεία να εξετάσουν πώς να γίνει δεκτή το έτοιμά μα. που είχαμε και στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου και στην Επιτροπή μας, έτοιμά μα λοιπόν για μεγαλύτερη κάλυψη των μεταναστών και των προσφύγων στο πλαίσιο της παιδείας ελπίζω να είναι πραγματικό το πρόγραμμα, δεν έχουμε περισσότερε λεπτομέρειε. Και μετά ανελήφθη κάποια υποχρέωση για να υλοποιηθεί καλύτερα η υλοποίηση των στόχων του 2020 και το Youth Report. Βέβαια δεν θέλω να σας πω κάτι άλλο. Αν πιστεύετε ότι μπορούμε ίσως να μοιράσουμε ένα σημείωμα για τους συναδέλφους που απουσίαζαν, ίσως ήταν καλό. Θεωρώ όμως η ιδέα μιας μια σχέση ως πιο στενής με τα εθνικά κοινοβούλια είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συνεχίσουμε. Σε αυτό το στάδιο θα ήθελα να ολοκληρώσω τις πληροφορίες που σας δίνω, να σας πω απλώς ότι έχουμε παρόντες, έχουμε μια ομάδα επισκεπτών που χαιρετίζω, εκεί στο βάθος κάθονται, 26 ακτιβιστές νέοι, πολιτικοί ακτιβιστές, από το Bulgarian Socialist Party. Προσκεκλημένοι συνάδελφο Μοντσενέκοφ, τους χαιρετίζω όλους και τους ευχαριστώ που παρακολουθούν ένα τμήμα των εργασιών μας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στη συζήτηση, μάλλον να περάσουμε στην έκθεση που πρέπει, ε, πρέπει να ψηφίσουμε. Έχουμε μεγάλο κατάλογο. Ας περάσουμε στην ψηφοφορία λοιπόν. Όσον αφορά την έκθεση Julie Ward, την ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά που έκανε για το ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, τη ποικιλομορφία ε, όσον αφορά τον πολιτισμό και την ε, παιδεία και τι θεμελιώδει αξίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάστηκε 21 Σεπτεμβρίου αυτή η έκθεση. 23 Οκτωβρίου ήταν η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Είχαμε 198 τροπολογίε. Λοιπόν, έγινε μεγάλη προσπάθεια και ευχαριστώ για, αυτούς και την, γι' αυτό και την γραμματεία για να καταλήξουμε σε συμβαστικέ προτάσει. Ευχαριστώ και του κοιόδη ηγητέ για τη δουλειά που έκαναν. Julie Ward, θα ήθελες να πεις δύο λόγια πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Έχεις το λόγο. Um, thank you very... Ευχαριστώ πολύ. Καθώς και τους κοιόδης και όλο το προσωπικό της γραμματείας αλλά και το δικό μου προσωπικό για όλα όσα έκαναν για αυτή την έκθεση. Επίσης τα δίκτυα οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ενδιαφέρθηκαν πολύ και έκαναν μια θετική συμβολή από πρακτικής απόψεως διότι εκείνοι αντιμετωπίζουν στην πράξη αυτά τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους. Νομίζω ότι αυξάνεται η ποιότητα των προσπαθειών και η σημασία του θέματος. Σας περάσουμε στην ψηφοφορία. Έχετε όλη την κάρτα για την ψηφοφορία. Παράγραφος 1, συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβίβα στική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 58 στην επόμενη σελίδα ίσως. Μαραγκάλ. Υπέρ τη 58 κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60. Σε δύο τμήματα είναι. Σε, με χωριστή ψηφοφορία είναι. Πρώτο τμήμα τη 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61 Ο κ. Χαλοντεύσκη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να συμπληρώσω το κείμενο της τροπολογίας 61. Υπογραμμίζει τη σημασία των έγκαιρων ε, μέτρων για την ενσωμάτωση κοινοτήτων οι οποίες είναι χωρισμένες. Συμφωνείτε όλοι, εντάξει. Όπως έχει τροποποιηθεί 61, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβα... Τροπολογία 100. Ναι. Υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίτ. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίτ. συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 σε δύο τμήματα. Θέλετε έλεγχο για την 115. Άρχεται για την 115 η ψηφοφορία επαλήθευσης. Πέρας. Δεν δουλεύει. Mm. Πέρας ψηφοφορίας.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 υπέρ πάλι κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 15 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 τροπολογία 130 υπέρ κατά αποχές έλεγχος 130 ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας Εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 142. Χωριστή ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά σε ελέγξουμε δεύτερο τμήμα της 142 έλεγχος πέρας εγκρίνεται συμβαστική 18 υπέρ κατά adopted we go to amendment 148 in favor in favor against abstention rejected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 20. Uh, hmm? Ακούτε. Ακούτε. 20, 20. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε νομίζω ότι εγκρίνεται Άρχεται η ψηφοφορία δεύτερο τμήμα της 29. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 30. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ με προφορική τροποποίηση ...37 υπέρ... ...κατά αποχές εγκρίνεται... ...συμβαστική 31 υπέρ... ...κατά αποχές εγκρίνεται... ...συμβαστική 33 υπέρ... ...κατά αποχές εγκρίνεται... Συμβαστική 33 υπέρ κατά αποχές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 με ε, ονομαστική κλίση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 23 υπέρ, 5 κατά και καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην Julie Ward. Και σε όλους βέβαια τους σκιώδεις εισηγητές. Τζούλι δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Ήταν πολύ σκληρή εργασία, ήταν όμως πολύ σημαντικά αυτά που πετύχαμε. Όταν ξεκινήσαμε πρώτα με την, για πρώτη φορά με την ιδέα αυτής της έκθεσης, αυτό ήταν πέρσι το καλοκαίρι και είχαν γίνει πολλά πράγματα έκτοτε, πολλά σημαντικά γεγονότα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι και οι συστάσεις της έκθεσης και οι διαβουλεύσεις που είχαν γίνει για την έκθεση αυτή απέκτησαν πολύ περισσότερη σημασία από ό,τι είχαν τότε. Αυτό που θα ήθελα να παροτρύνω όλα τα μέλη της ε, Επιτροπής μας να κάνουν είναι να φέρουν αυτή την έκθεση στα κράτη-μέλη τους στις, ε, στους αρμόδιους για την παιδεία <clears throat> και την νεότητα γιατί αυτή η έκθεση πρέπει να εφαρμοστεί θα πρέπει να δημιουργηθεί κάποια εμπιστοσύνη στους πολίτες μετά από όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει και να ενισχυθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος επί τη βάση αυτού που θεωρήσαμε όλοι ότι είναι οι βέλτιστες πρακτικές. Πρέπει να το κάνουμε αυτό γιατί είναι υποκίνδυνο οι θεμελιώδεις αρχές μας και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ζούμε σε μια συνεκτική και ειρηνική κοινωνία όπου οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν ειρηνικά. Ευχαριστώ Τζούλη και για αυτή την ε, όθηση που έδωσε. Είναι σημαντική αυτή τη στιγμή. Είναι στρατηγική σημασία να μιλάμε για αυτά τα θέματα στην Ευρώπη και στι χώρε μα. Α, συγγνώμη. Σημαντική στρατηγική σημεία, λέει εγκλειστή η πρόεδρο. Και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο κουβεντιάζονται. Θε να προσθέσει κάτι. Να ζητήσω συγγνώμη που δεν μπορώ να μείνω στη συνεδρίαση. Είμαι πολύ ενεργό μέλος της Επιτροπής ήταν εργασία μια ζωή ο πολιτισμό και η παιδεία. Αλλά οι εκλογές μας στη βορειοδυτική Αγγλία έχουν πρόβλημα. Έγιναν πλημμύρε το Σαββατοκυριακό. Και είμαι η μόνη ευρωβουλευτή που είμαι στην επαρχία της Κάμπρια που έγιναν, συνέβησαν οι πλημμύρες. Έχω πολλές κατεπίγους καταστάσεις να αντιμετωπίσω παρόλο που είμαι εδώ αυτή την εβδομάδα. Θα έμενα γιατί με νοιάζει το πρόγραμμα που συζητούμε, αλλά για την ώρα πρέπει να φύγω. Ελπίζω να με συγχωρέσετε γι' αυτό. Βεβαίως, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας για τη Βορειοδυτική Αγγλία. Ευχαριστώ να υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει τον Μάρτιο της εκθέσεως αυτής και μετά πάμε τώρα στη συνέχεια του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία όσον αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη 2020 εισηγητής είναι ο κύριος Κρασνοτζεύσκη τον ευχαριστώ για την παρουσία του α δεν τον έβλεπα Ξέρουμε απόλυτα πως αυτό το ζήτημα για μας είναι στρατηγική σημασία και υπό το φως όλων αυτών που συμβαίνουν και συνέβησαν θα πρέπει να δούμε κατά πόσο οι προτεραιότητες ε, που ετέθησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνονται αποδεκτές ή πρέπει να ισχύσουμε κάποιες στρατηγικές και μετά από αυτά που ακούσαμε στη διακοινωνιστική ε, διάσκεψη θα πρέπει να αποτιμήσουμε, να λάβουμε υπόψη αυτά που ακούσαμε από τους νέους, να τα λάβουμε υπόψη και βέβαια και να εκφράσουμε και δικές μας σκέψεις. Ο εισηγητής θα παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής του στην επόμενη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου, 17-18 Φεβρουαρίου, ψηφοφορία θα γίνει τον Απρίλιο. Λοιπόν, έχουμε χρόνο, έχουμε δυνατότητα μιας πρώτης ανταλλαγής ε, απόψεων σήμερα. Θα δώσω σε εσά, αγαπητέ εισηγητά, κύριε Κρασνοδιέσκη, το λόγο. το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρουσιάσω μερικές από τις κυριότερες ιδέες που σκέφτηκα διαβάζοντας αυτή την έκθεση. Βεβαίως το θέμα είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε σοβαρά, αλλά δεν θέλησα να γράψω μια έκθεση όπου θα εκθέτουμε μόνο καλές προθέσεις. Διότι σε άλλες, και σε άλλες εκθέσεις έχουμε εκφράσει επικρίσεις και λήψεις για αυτούς που φεύγουν νωρίς από το σχολείο ας πούμε. Λυπόμαστε γιατί αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται η αγραμματοσύνη, ο αναλφαβητισμός. Θελήσαμε λοιπόν να τονίσουμε τη στρατηγική του 2020 διότι φυσικά αυτό που θέλουμε είναι να δούμε κριτικά το πρόγραμμα και επειδή σήμερα είναι περιορισμένος ο χρόνος μας θα ήθελα να τονίσω τρία κύρια θέματα αλλά βέβαια μπορώ να αναλάβω και να ακούσω και ό,τι σχόλιο έχετε άλλο. Πρώτον, θα εξετάσω την οργανωτική δομή του προγράμματος και τους διάφορους τομείς που αναφέραμε και προηγουμένως. Φυσικά προβλέπονται αλλαγές και το Κοινοβούλιο τις έχει αναλύσει πολλές φορές. Αυτά αποφασίζονται από τις ομάδες εργασίας, διότι μια νέα διαδικασία με την βάση την οποία ιδρύθηκαν αυτές οι ομάδες εργασίας προβλέπει η σύνθεσή τους να διευρυνθεί, να αλλάξει διότι η παιδεία είναι κάτι σημαντικό και διότι υπάρχει το σοβαρό θέμα ας πούμε της σύνδεσης μεταξύ οικογενειακής ζωής και σχολικής τι αυτής. Δεν έχουμε μέχρι σήμερα πει τίποτα για το ρόλο των γονέων ούτε έχουν έρθει εκπρόσωποι των γονέων για διαβούλευση. Το θέμα είναι πολύπλοκο ίσως στη φύση του, διότι δίνουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε ποσοτικούς δείκτες. Πρέπει να τονίσουμε λίγο περισσότερο την ποιότητα. Ξέρω ότι η ποιότητα είναι δύσκολο να μετρηθεί και να αξιολογηθεί, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι πολύ εύκολο να κάνουμε στατιστικούς πίνακες με βάση ποσοτικές αλλαγές και να έχουμε ποσοτικούς δείκτες. Αλλά σε πολλές χώρες, παρά το ότι βελτιώνονται οι δείκτες, εγώ ξέρω τον τομέα της παιδείας γιατί ήμουν δάσκαλος πολλά χρόνια, ξέρουμε ότι τα στατιστικά στοιχεία δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στην πραγματικότητα. Και ίσως λοιπόν να έπρεπε να το ξανασκεφτούμε αυτό. Και τα εκπαιδευτικά συστήματα να τονίζουν λίγο παραπάνω την εκμάθηση δεξιοτήτων. Εκπαιδευτικά συστήματα δηλαδή βασισμένα σε πραγματική γνώση. Ξέρουμε ότι συχνά ακούγεται αυτή η έμφαση που θέλουμε να δώσουμε στην απόκτηση δεξιοτήτων αλλά καμιά φορά αυτό καταλήγει να παραγνωρίζει την απόκτηση των βασικών γνώσεων. Δεύτερον, θα τονίσω την ποιότητα της παιδείας και τη σύνδεση μεταξύ της ποιότητας της παιδείας και της αγοράς εργασίας διότι προφανώς αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι να σπουδάσουν με ανώτερη εκπαίδευση 25% των αποφύτων σχολείων ξέρουμε ότι δεν αποκτούν περισσότερες διπλώματα. Επίσης θέματα που αφορούν τη διαδικασία της Μπολόνιας. Φαίνεται ότι υπάρχει εδώ ένα χάσμα μεταξύ των αξιολογήσεων που έγιναν του προγράμματος και από την άλλη μεριά εκείνων που ωφελούνται από αυτό. Άλλη άποψη έχουν αυτοί. Και ένα από τα στοιχεία νομίζω που πάντα επικρίνονται είναι ό,τι αφορά τον κατακαιρματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Βεβαίως υπάρχουν και θετικές πλευρές στη διαδικασία της Βολονίας. Αλλά υπάρχουν ένα-δυο στοιχεία που με κάνουν διστακτικό. Σαν να βλέπω δηλαδή εδώ μια προειδοποίηση, αυξάνεται η γραφειοκρατία ας πούμε σε σχέση με τη διαδικασία αυτή. Γι' αυτό θα εξετάσω και αυτό το θέμα. Και με χαρά θα ακούσω αν έχετε σχόλια. Και το τρίτο μέρος, η τρίτη ιδέα της εκθεσής μου θα βασιστεί σε κάτι που και εσείς η ίδια κυρία Πρόεδρε είπατε. Έχω ένα χρονίζον πρόβλημα γιατί μιλάμε για την εκπαίδευση όχι μόνο παιδιών αλλά και ενηλίκων και μεταναστών. Σήμερα είναι ιδιαίτερα κέριο αυτό το πρόβλημα βέβαια γιατί ξέρουμε ότι το όλο θέμα της μετανάστευσης γίνεται όλο και σπουδαιότερο. Έρχονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική αλλά υπάρχει και ενδοευρωπαϊκή μετανάστευση οι μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά των μεταναστών έχουν περισσότερα προβλήματα από τα υπόλοιπα στην παιδεία και ίσως και οι ίδιοι οι ενήλικες. Η επαγγελματική τους εκπαίδευση είναι πιο δύσκολη από των υπολείπων. Και στην έκθεση που μόλις συγκρίναμε γινόταν λόγος για διαπολιτιστικό ή διαπολιτισμικό διάλογο για να υπάρξει καλύτερη συμπερίληψη και των μεταλλαστών στην εθνική ζωή. Κάμια φορά οι μετανάστες βέβαια έρχονται για λίγο χρόνο στην Ευρώπη και κερδίζουν ορισμένα χρήματα και μετά ξαναφεύγουν αλλά υπάρχουν και άλλοι που μένουν περισσότερο και πρέπει να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση για αυτούς και ως προς την εθνική κληρονομιά της κάθε χώρας. Πρέπει να αυξηθεί η συνεργασία διότι μερικές χώρες έχουν περισσότερη πείρα στον τομέα αυτών από άλλες. Αυτά είναι οι τρεις κύριες ιδέες στις οποίες θα βασιστώ τα τρία κυρία θέματα αν θέλετε και ελπίζω και εσείς κυρίες και κύριοι να δεχτείτε αυτή τη γενικότερη δομή που προτείνω και ό,τι σχόλια έχετε προφανώς θα με βοηθήσουν να επανεξετάσω πληρέστερα μερικές από αυτές τις ιδέες. Αλλά θέλω να κρατήσω μια συνέπεια στη, στο κείμενό μου δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα από την αρχή σε μια έκθεση αλλά νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να προετοιμάσουμε έγγραφο έκθεση που να εκφράζει τις ευχές μας αλλά και την πραγματικότητα. Αυτό θέλω να κάνω. Ρεαλιστική έκθεση. Σας ευχαριστώ κύριε Κρασνογεύση. Συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί να εστιαστούμε σωστά, να κάνουμε προτάσεις και να επανεξετάσουμε τις προτεραιότητες. Είναι πολύ σημαντικό. Από τη δουλειά σας απορρέει αυτό, από τη συνεργασία με τους κοιώδεις και από τις εργασίες επιτροπής. Και αναφορά στην ποιότητα των δικτών. Οι ποιοτικοί δείκτες είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Τι θα ήθελα να κάνω. Έχουμε 30 λεπτά για ερωταπαντήσεις για να τηρήσουμε το χρόνο. Πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές που είναι παρόντος και μετά στους άλλους συναδέλφους που θα στείλει το λόγο. Μετά θα δώσουμε το λόγο στους συντονιστές βέβαια. Οι συντονιστες δυο δύο-τρία λεπτά παρόλο που είναι λίγοι παρόντες. Και μετά τα άλλα μέλη ένα-δύο λεπτά. Σύντομα δηλαδή. Οι σκιώδεις πρώτα απ' όλα που θέλουν να πάρουν το λόγο, μετά οι συντονιστές. Ορίστε. Σέντροβα. Ένα, δύο, τρει, τέσσερι έχω που ζήτησαν πέντε συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη ζητώ γιατί θα χρειαστεί να φύγω γιατί είμαι συγγήτρια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Απασχόληση. Θα ξαναγυρίσω όμως η έκθεση του κυρίου Τέσκι νομίζω ότι γενικά με βρίσκει σύμφωνη. Με βρίσκει σύμφωνη η δομή της, με βρίσκει σύμφωνη το γεγονός ότι πρέπει να δούμε και το ποσοτικό και όχι μοναχα το ποιοτικό τμήμα της παιδείας. Οι ποιοτικοί δείκτες τώρα θα πρέπει να τύχουν προτεραιότητα σε ορισμένους τομείς ιδίως όταν τα προγράμματα αυτά θέλουν να βελτιώσουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων την, στην, στην παιδεία. Όταν ε, είδαμε την παρουσίαση της Κομισιόν ήταν εφανερό ότι υπάρχει βελτίωση της ποιότητας. Φυσικά αυτό εξαρτάται από τους τομείς, αλλά γενικά υπάρχει βελτίωση της ε, ποιότητας. Εγώ θέλω να εστιάσω περισσότερο στην προσχολική εκπαίδευση, η οποία έχει σημαντική επίπτωση γενικά στην ποιότητα της παιδείας. Θα πρέπει εκεί να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα και όχι μόνο στην ποσότητα της παιδείας. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα στην προσχολική εκπαίδευση. Αυτό προφανώς είναι πιο δύσκολο να το καταμετρήσει κανείς. Και η αξιολόγηση ως εργαλείο Βελτίωση των αποτελεσμάτων υπό το πρίσμα της ποιότητας είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να θεωρηθεί τμήμα του πλαισίου μας. Τώρα το θέμα της ενσωμάτωσης διαφόρων κοινοτήτων, αυτό είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Είναι πολύ σημαντικό να επεκταθούμε περισσότερο στον χώρο αυτό. Κάτι το οποίο θα ήθελα να αναφέρω και ίσως θα μπορούσε να διευκρινιστεί καλύτερα είναι η παιδεία σε ό,τι αφορά τα τις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. Και είναι σημαντικό αυτό να το δούμε όχι μόνο χάσαμε μια προσωπική υπόθεση των μαθητών, αλλά και μια ανάγκη ενσωμάτωσης των νέων μαθητών που έρχονται στα σχολεία ως μετανάστες. Επίσης υπάρχει η λεγόμενη ηθική διαπαιδαγώγηση και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ που είστε το χρόνο. Συνάδελφε Μαραγκάλ, έχετε το λόγο. Μαργκάλ. Ζητήσατε το λόγο. Ευχαριστώ. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να επεξεργαστούμε αυτή την έκθεση, να τη διαβάσουμε και με μεγάλη προσοχή πρώτα. Ελπίζω ότι θα έχω στο μέλλον την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις και με τον εισηγητή. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω τώρα και είναι το εξής τα εκπαιδευτικά μας συστήματα στην Ευρώπη, τουλάχιστον στο πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο, βρίσκονται πολύ μακριά από το να θεωρηθούν ευρωπαϊκά συστήματα. Εθνικά συστήματα, φυσικά σε πολλές περιπτώσεις είναι απόλυτα αξιόπιστα, σε πολλές περιπτώσεις όμως <clears throat> έχουν ελλείψεις σε ό,τι αφορά την ε, παιδεία για την ε, Ευρώπη και έχουν μια υπερβολική εσωστρέφεια. Θα ήταν λοιπόν πολύ χρήσιμο να θέσουμε αυτά τα συστήματα τα εκπαιδευτικά σε μεγαλύτερη επαφή μεταξύ τους. Δεν ζητώ η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιομιστεί τις αρμοδιότητες για τα θέματα παιδείας. Αυτό θα ήταν παράλογο. Αλλά υπάρχει ένα σημαντικό έδαφος για να μπορέσουμε να προωθήσουμε περισσότερο μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα που έχουν να κάνουν με τις άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί κανείς μέσα σε αυτές τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα με ραγδαίο ρυθμό να παραμείνει μέσα στο καβούκι του. και στην ε, ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση έχουμε το σύστημα της Μπολόνιας και έχουμε και το σύστημα, του, το σύστημα Έρασμος. Είναι δύο θετικά στοιχεία και τα δύο, αλλά στο δευτεροβάθμιο επίπεδο δεν έχουμε κανένα σύστημα ανταλλαγής ή κάποιο σύστημα μηδέας αναγνώρισης, ούτε Μπολόνια ούτε Έρασμο. Πρέπει να βρούμε λοιπόν κάποια συστήματα τα οποία θα μας επιτρέπουν να έχουμε μια καλύτερη βαθμονόμηση, αμοιβαία αναγνώριση και <clears throat> αποτίμηση του επίπεδου ποιότητος, καλύτερη αποτίμηση του επίπεδου εκπαίδευσης των διδασκόντων. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε προσθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με επικοδομητικό τρόπο, αυτό θα είναι πολύ χρήσιμο να δώσουμε και περαιτέρω δυνατότητες μάθησης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ νομίζω ότι βρίσκεται ο πυρήνας που θα πρέπει να είναι το θέμα που μας απασχολεί περισσότερο σε αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστώ. τα αυτά που υπογραμμίσατε, συμφωνώ μαζί σας. Λιμπάτσκα, συνάδελφε Λιμπάτσκα. Ευχαριστώ. Έχω ένα-δύο σχόλια και κάποιες παρατηρήσεις, αν επιτρέπει ο κύριος Κναστοντιέψκη. Δεν θα ήθελα να στιαστώ μόνο στους ποιοτικού δείκτες, αλλά και στους επίσημους δείκτες. Δεν είναι μόνο θέμα ποιότητας, διότι καμιά φορά δεν έχεις πολύ καλούς επίσημους δείκτες, οπότε δεν έχεις καλή γενική εικόνα. Ο κ. Κασνοντέψκι αναφέρθηκε στην εκπροσώπηση των συλλόγων γονέων στις ομάδες εργασίας. Έχουμε τους μαθητές, τους διδασκάλους και τους γονείς. Αυτό το τρίγωνο έχουμε σε σχολικό επίπεδο. Οπότε θα έπρεπε να έχουμε και σωστή εκπροσώπηση και σε αυτό το επίπεδο. Τώρα η διαδικασία της Μπολόνια ένα θα σας παρότρινα να κάνετε. Να μην αναμειγνύουμε τη διαδικασία της Μπολόνια με την αξιολόγηση. Είναι διαφορετικά πράγματα. Πολλά θα πρέπει να κάνουμε ούτω ώστε να προσαρμόσουμε τη διαδικασία της Μπολόνια για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού ακαδημαϊκού χώρου. Προφανώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό ε, με κάποιο πετυχημένο πρόγραμμα. Τέλος, δεν ξέρω αν και ο Κρασνοντέψκι θα ήθελε να το κάνει ή ήθελα να το παραλείψει. Δεν λέμε αρκετά όσον αφορά τις αλλαγές νοοτροπίας παραδείγματος αν θέλετε προτύπων που έχουμε στα σχολικά προγράμματα για να εργάζονται οι νέοι στην αγορά εργασίας και να βρίσκουν ε, θέσεις εργασίας στο σύγχρονο κόσμο. Θα πρέπει να αλλάξουμε τα πλαίσια θα πρέπει να έχουμε πιο δημιουργικές καινοτόμες μορφές εκπαίδευσης διότι τίθεται θέμα δεξιοτήτων, πολιτισμικών κωδίκων κλπ. Αλλά όταν μιλάμε για την ανάγκη για παιδεία, για κατάρτιση, θα πρέπει να πούμε ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα είναι υπεύθυνα για την ε, ποιότητα προετοιμασία των νέων, τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζουμε του νέου για την αγορά εργασία. Το σύστημα όμω αυτό δεν είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Οπότε έχουμε δύο έννοιε, δύο ιδέε που δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται. Δεν μπορεί να περιμένει κανεί από εμά να βρούμε τη μαγική συνταγή, ούτω ώστε ο κάθε νέο να βρίσκει δουλειά. Θα πρέπει να εκπαιδεύουμε, να καταρτίζουμε τον κόσμο, να προσπαθήσουμε να καλύψουμε τι ανάγκε τη αγορά-εργασία, αλλά όχι και απαραίτητα να δημιουργούμε θέσει εργασία. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Ευχαριστώ, συνάδελφε Λιμπάτσκα για αυτά που υπογραμμίσατε. Ο κύριος Χουντής έχει το λόγο. Ορίστε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι νέο μέλος στην Επιτροπή και επομένως αν έχει ξανασυζητηθεί το θέμα ε, συγχωρέστε με δεν το άκουσα αλλά ε, επειδή θέλω να είμαι ενεργό μέλος της Επιτροπής ακούγοντας τον εισηγητή σε αυτά τα κρίσιμα θέματα που θέλει να δουλέψει στην έκθεσή του και βεβαίως προετοιμαζόμενος διάβασα την απόφαση του Συμβουλίου για τα θέματα αυτά ε, του Μαΐου του 2009 θα πω ορισμένες σκέψεις ίσως και με τη μορφή ερωτημάτων ε, και στην τελική διατύπωση θα πω και τις απόψεις μου για τα θέματα που πρέπει να έχει έκθεση. Ερώτηση πρώτη. τι εξετάζουμε, τι θέλουμε να εξετάσουμε. Την κατάσταση της παιδείας, της εκπαίδευσης και τον συντονισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλιστα. Μπαίνουν κάποιες προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες αυτές έχουν τεθεί με τη σημερινή πραγματικότητα ή στη βάση των προτεραιοτήτων και των στόχων της, στρατηγική της στρατηγικής της Λισαβόνας η στρατηγική της Λισαβόνας γνωρίζετε αγαπητοί συνάδελφοι, επεξεργάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2000, απέτυχε, απέτυχε και ως πρώην Ευρωβουλευτής στην προηγούμενη διάστημα δεν είχε γίνει ποτέ μια αξιολόγηση. Πού πήγε ο στόχος για την πλήρη απασχόληση, πού πήγε ο στόχος ότι η Ευρώπη θα είναι η πιο ανταγωνιστική οικονομία του κόσμου το 2010. Πάμε όμως παρακάτω. Δεν θα το λύσει η έκθεση αυτό. Στη συνέχεια έχουμε τη στρατηγική 20, 20, Εκεί λοιπόν αυτά έγιναν μεσούσεις της οικονομικής κρίσης. Η οικονομική κρίση είχε συνέπειες και στα ζητήματα της παιδείας, της εκπαίδευσης, θα πω δύο-τρία στοιχεία. Ιδιαίτερα σε ορισμένες χώρες. Επομένως η δεύτερη ερώτηση είναι η έκθεση ε, τα αποτυπώνει αυτά ως θέματα. Τρίτη πλευρά. Η κρίση είχε ε, έχει, είχε δραματικές εξελίξεις και στον τομέα της παιδείας, ιδιαίτερα σε ορισμένες χώρες, ειδικά στη χώρα μου την Ελλάδα. Δύο συμπτώματα θα σας πω, αφού συζητάμε την ποιότητα. Το πρώτο, περικοπές στη δημόσια εκπαίδευση, με συνέπεια να υπολειτουργούν πανεπιστήμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και τα άλλα επίπεδα. Και δεύτερο, που έχει σχέση με την ποιότητα, ο συνάδελφος επειδή άκουσα ότι είναι εκπαιδευτικό, θα το καταλάβει καλύτερα και εμεί θα το καταλάβουμε καλύτερα όσοι έχουν περάσει μέχρι στιγμή. Γερνάει, δηλαδή μεγαλώνει ο μέσο όρο τη ηλικία των εκπαιδευτικών, καθώ δεν διορίζονται καινούργοι. Και ξέρω ότι αυτό το φαινόμενο υπάρχει και σε άλλε χώρε, λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών. Αυτό, ναι, το, το, το έχω κουβεντιάσει και με άλλου συναδέλφου και είναι ένα πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό θα το θίξουμε ω θέμα ποιότητα τη παιδείας Δηλαδή εκπαιδευτικό προσωπικό, χαμηλός χρηματοδοτικό, χρηματοδότηση και ούτω καθεξής. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, γιατί με την επιφύλαξη, αλλά με την υπογράμμιση ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, είναι πάρα πολύ, και με την υπόσχεση που έδωσε ο εισηγητής μας και την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όλοι, να αποτυπώσουμε πράγματι, την πραγματικότητα σήμερα σε αυτό το θέμα. Και μια τελευταία ηρωνική, ηρωνική ομολογώ, παρατήρηση. Αν το 2009 ή πριν μιλούσαμε για συντονισμό στην εκπαίδευση στις χώρες της Ευρώπης και το αποτέλεσμα, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως το γνωρίζετε πολύ καλά ή ενδεχομένω αν δεν το γνωρίσετε να σας το πω, είναι να φεύγουν από τις χώρες του Νότου επιστήμονες με πτυχία, με τα πτυχιακά και να πηγαίνουν, πηγαίνουν στις χώρες του Βορρά και αυτό ηρωνικά ξαναλέω, να θεωρείτε ότι επιτεύχθηκε ο συντονισμός δεν νομίζω ότι πρόκειται περί αυτού. Αν δηλαδή τα καλύτερα μυαλά, του εκπαιδευμένου ανθρώπου, λόγω των οικονομικών και άλλων δυσκολιών, φεύγουν και πάνε στι βορειότερε χώρε, δεν έχουμε συντονισμό. Επομένω, ε, νομίζω ότι πρέπει να το δούμε με βάση την πραγματικότητα. Είναι φιλόδοξη η έκθεση. Ε, συγχωρέστε με αν είπα κάτι παραπάνω που το έχετε κουβεντιάσει, αλλά ε, υπόσχομαι όταν θα διαβάσουμε την έκθεση και με τι παρατηρήσει όλων να την κάνω καλύτερη ή να προσπαθήσω να σα πω κι εγώ πιο συγκεκριμένα ποιε θα ήταν οι δικέ μου παρατηρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε αντιθέτω για αυτή τη σημαντική παρέμβασή σα. Νομίζω ότι είναι πολύτιμο να βλέπουμε διαφορετικέ προσεγγίσει και να υπάρχουν και συγκεκριμένε προτάσει που θα κάνουμε. Είναι σαφέ ότι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να δούμε είναι να επαναπροωθήσουμε τον κεντρικό χαρακτήρα των επενδύσεων που δεν είναι κόστος, είναι επενδύσεις για την παιδεία και την εκπαίδευση. Συνάδελφε Μόργανο, ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ αντιδρώ σχετικά με την εισαγωγή του συγκητού και θα ήθελα όμως να δω και ένα έγγραφο, ένα κείμενο για να μπορώ να κάνω συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω κάποια θάματα προσπαθώντας να μην επαναλαμβάνω τα υποθέντα από τους συναδέλφους. Ε, συμφωνώ όσον αφορά ότι χρειάζεται να εστιαστούμε επί κάποιων ζητημάτων, ε, να μην καλύπτουμε τα πάντα, διότι σαν Επιτροπή μπορούμε να δείξουμε ικανότητες, να εντοπίζουμε προτεραιότητες σε σχέση με το συνολικό θέμα. Δεύτερο, πιστεύω ότι όταν μιλάμε για ποιότητα σήμερα απαιτείται και κάτι παραπάνω να δείξουμε. Δηλαδή να μπορέσουμε να υπογραμμίσουμε κάποια διέξοδο πρέπει να την καθορίσω καλύτερα για να μην μιλάω γενικόλογα. Όπως αυτά που μας είπε ο εισηγητής. Θέλουμε μια θέση και αντιπαράθεση σε σχέση με δείκτες και ποιότητα. Να εξετάσουμε τους ποιοτικούς δείκτες. Όχι όλους, να δούμε τους δείκτες εκείνους που θεωρούμε ότι θα πρέπει ε, να είναι σωστοί για να μην επαναληφθούν ήδη παρελθόντα προβλήματα όσον αφορά τις προοπτικές που υπάρχουν. Συμφωνώ με αυτά που ήδη τονίστηκαν. Ξέρουμε πολύ καλά τις αρμοδιότητες, πολύ περιορισμένες Ευρωπαϊκής Ενώσης στον τομέα. Μπορούμε όμως να ασκήσουμε πιέσεις για να υπάρχει ένας κάποιος συντονισμός των διαφόρων συστημάτων, των εκπαιδευτικών, σε διάφορα επίπεδα. Ανωτάτη εκπαίδευση, πανεπιστημιακό επίπεδο, κάποιοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στη δικασία της Βολόνια και στη Λισαβόνα, συνθήκη Λισαβόνας. Εγώ δεν θέλω να επαναλάβω αυτά. Θα επέμενω όμω το κείμενο στο να τονίσουμε τη βασική κατάρτιση και εκπαίδευση. Και το λέω αυτό αναφερόμενος και στην, στην ε, παιδεία για την ευρωπαϊκή ευθυγένεια. Ένα πολιτική πολιτικής αγωγής που χρειάζεται. Δηλαδή ε, ζούμε σε ένα πλαίσιο που διατρέχουμε κάποιου κινδύνου. κινδύνους. Άθελά μα και το λέω προκλητικά αυτό, αποκλειστικά να βασιστούμε στην ιδέα ε, της προσέγγισης βασιζόμενη μόνο στην αγορά εργασίας και ξέρουμε ότι η αγορά εργασίας σήμερα δεν δίνει εχέγγυα όσον αφορά τις γνώσεις. Πρέπει να υπάρχει σεκτισμός παιδείας παραγωγικών συστημάτων. Υπάρχουν 2 με τρεις χιλιάδες νέα επαγγέλματα που δεν ξέρουμε πολύ καλά και είναι ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και ποιο θα είναι το περιεχόμενο των νέων θέσεων. Ε, θα ήθελα να έχουμε ένα τέταρτο τμήμα, όπως ανέφερθηκε από τον συνάδελφο Λιμπάσκα. Να αναφερθούμε στις αλλαγές που ξεκίνησαν και λαμβάνουν χώρα και αφορούν και το μέλλον. Σήμερα όποιος ξεκινά την εκπαίδευση, όταν τελειώνει την εκπαίδευση, ίσως τελικά να βρεθεί εκτός νυμφώνος, δηλαδή εκτός των σχέσεων με την αγορά εργασία και κάτι άλλο που ανέφερε ο συνάδελφος Σιντρόβα που εξήλθε να αναφερθούμε και στα προσχολικά θέματα. Έγινε αναφορά και στη Λισαβόνα πάνω σε αυτό. Είναι νομίζω σημαντικό στο σφαιρικό πλαίσιο που συζητούμε. Πρέπει να πείσουμε ότι ό,τι γίνεται στα πλαίσια της κατάρτισης και της παιδείας είναι μια επένδυση. Δεν είναι απλώς δαπάνη, όπως καμιά φορά αναφέρεται και συνεχώς επαναλαμβάνεται αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσω το λόγο. Αν θα θέλανε να προσθέσουν κάτι πλέον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστώ που είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. πολύ κύριε Πρόεδρε και για την ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Και εμεί είχαμε μια πολύ θετική συζήτηση με τον εισηγητή κύριο πριν από τη συνεδρίαση αυτή για πολλές πτυχές της έκθεσης και νομίζω ότι σήμερα θα ήθελα να τονίσω απλώς την ομορφιά του πλαισίου αυτού, την ωραιότητα την προτεραιότητα που θέλουμε να δώσουμε σε όλα τα επίπεδα της παιδείας πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και όλους τους τύπους μάθησης μιλάμε και για την επίσημη παιδεία και για την άτυπη είναι λοιπόν ε, η έκθεση αυτή με ένα πρώτο βήμα συνεργασίας με το Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη και μας για να προωθήσουμε αυτές τις προτεραιότητες. Επίσης είναι σημαντικό ότι ακούγοντας αυτά που είπατε καταλαβαίνω ότι το γενικότερο πλαίσιο που προβλέπουμε μπορεί να συμπεριλάβει πολλά από αυτά που είπατε την εξισορρόπηση μεταξύ παιδείας και απασχολησιμότητας, απόκτησης δεξιοτήτων, το λέει ρητά αυτό η έκθεση και απ' την άλλη επίσης ο σημαντικός στόχος της ε, των πολιτών και στην αγωγή του πολίτου, στην συμπερίληψη όλων στις κοινέ αξίες. Αυτές οι δύο προτεραιότητες εξισορροπούνται εδώ πολύ ωραία. Επίσης ξέρουμε ότι και η ανακοίνωση είχε θελήσει να συμπεριλάβει αυτές τις προτεραιότητες στο πρόγραμμα εργασιών της Κομισιόν και ιδιαίτερα αυτά που υπέγραψαν οι Υπουργοί Παιδείας το Μάρτιο ως συνέχεια στις επιθέσεις κατά του Αρλί Εμπντό. Μία δήλωση δηλαδή να προωθηθούν περισσότερο οι κοινέ αξίες μέσω της παιδείας. Και αυτό επίσης ανταποκρίνεται συμπεριλαμβάνεται πλήρως στο σχέδιο της έκθεσης ή προσχέδιο. Κάτι άλλο τώρα για τις επενδύσεις. Βλέπετε ότι μεταξύ των προτεραιοτήτων είναι η πλήρης χρήση του ε, επενδυτικού σχεδίου μαζί με την ΕΤΕ διότι γνωρίζουμε ότι έχουν υπάρξει περικοπές στους προπολογισμούς της παιδείας. Για την προσχολική ηλικία η Κομισιόν συμφωνεί με όσους τόνισαν τη σημασία της γιατί υπάρχουν πολλά στοιχεία για τον σημαντικό ρόλο που θα έπαιζε μία αρχή, μία εκπαίδευση νωρίς. Και τέλος αυτά που υπόθηκαν για τους δείκτες συζητήσαμε με προσώπους των χωρών μελών για τους τωρινούς δείκτες και benchmark και δεν ζήτησε κανείς ε, αλλαγές. Ξέρουμε ότι είναι ποσοτικοί και ότι δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα αλλά κανείς δεν και εγώ να τους αλλάξει. Φυσικά και εμείς συμφωνούμε ότι χρειάζονται περισσότεροι ποιοτικοί δείκτες Παρ' όλα αυτά ξέρω ότι θα έχετε μια παρουσίαση και από συναδέλφους μας στην Κομισιόν όπου θα δείτε και μια πιο ποιοτική ανάλυση μαζί με την ποσοτική. Ελπίζω να μην μακρηγόρησα. Σας ευχαριστώ μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσω. Όχι, σας ευχαριστώ πραγματικά κυρία Σοφία Έριξον για την παρέμβασή σας. Αντιθέτως, χρησιμότατη για τη συζήτησή μας. Πιστεύω ότι δεν θέλω να επαναλάβω τίποτα από τα υποθέτα, αλλά να προσθέσω δύο στοιχεία. Να αξιολογήσουμε κάθε δύο πτυχές, θα έλεγα. Αύξηση κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη σε σχέση με την πρόσβαση και τη συνέχεια των σπουδών. Δεν θα ήθελα να είναι εκτό πλαισίου αυτό. Η κρίση κλπ. Πιθανότατα είναι ένα άλλο θέμα, ότι το σχολείο δεν είναι πλέον σαν κοινωνικός ανελκυστήρας όπως ήταν αλλά είναι ένα στοιχείο επενδύσεως στις μελλοντικέ γενιές. Θα πρέπει να τεθεί το θέμα και στα πλαίσια τα ευρωπαϊκά. Να έχουμε επίγνωση ότι καμιά φορά και την πρόσβαση στα προγράμματα κινητικότητας αυτό παίζει ρόλο. Το είδαμε και στο Youth Forum. Με ευχαριστεί ότι, επανεξ... ότι εξισορροπήθηκε και άτυπα και επίσημα και το θέμα της ευρωπαϊκής ηθαγένειας, ενεργού ηθαγένειας που έχει τεθεί. Μετά θα πρέπει να καλέσουμε και τα κράτη-μέλη να φροντίσουν για τα εκπαιδευτικά συστήματα και την κυβέρνηση αυτών, να υπάρχει μια προσέγγιση, αν θέλετε, των συστημάτων αυτών. Να υπάρχει προσέγγιση αν φάση τι και τη βαθμολόγηση benchmark. Ίσως θα ήταν σημαντικό, εφόσον συζητούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δούμε πώς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ΕΦΣΙ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε επενδύσεις για την παιδεία. Θα είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε, αλλά ίσως μπορούσαμε ήδη να το θίξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας. Θέλει να πει κάτι ο εισηγητής, ο κύριος Κρασνοντεύσκη. Ε, ε, Συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τα σχόλιά σας και βλέπω στην περαιτέρω συζήτηση μαζί σας όταν υπάρχει η γραπτή μορφή της έκθεσης. Είχαμε ήδη μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ακούσαμε και την άποψη της Κομισιόν. Έχετε δίκιο, είναι πολύ καλό το πρόγραμμα αυτό, είναι ιδιαίτερα ελκυστικό ιδίω όταν μπορούμε να συνεργαστούμε μεταξύ μας και να εξασφαλίσουμε τον ε, σεβασμό για όλες τις εθνοτικές ομάδες. Βέβαια ξέρουμε ότι υπάρχει πολυμορφία στα συστήματά μας, αλλά τα συστήματά μας έχουν τις ίδιες αρχές. Να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους και να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζονται και στην αγορά εργασίας. Τώρα μέχρι που θα το φτάσουμε αυτό, χρειάζεται πραγματισμός. Αλλά δεν θέλουμε να εκπαιδεύουμε μονάχα χειρονάκτες, δεν θέλουμε να εξάγουμε τους επιστήμονές μας, θέλουμε να έχουμε λοιπόν παιδεία αλλά υπάρχει παράλληλα και ο στόχος της προσαρμογής προς την ε, ε, αγορά. Θέλουμε οι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε στα πανεπιστήμια να μπορέσουν να είναι και πολίτες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι. Δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε μόνο κομφορμιστές, θέλουμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα μεγάλο φάσμα δεξιοτήτων και απόψεων και θέλουμε να έχουν αυτοί οι άνθρωποι και αστική συνείδηση ως πολίτες και να έχουν θάρρος σε σχέση με τα θέματα αυτά. Κάποιοι λοιπόν δεν τελειώνουν ποτέ την παιδεία τους. Επομένως δεν είναι μοναχα θέμα παιδείας, είναι θέμα του να καταλάβουμε και την ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Όλα αυτά είναι σημαντικά λοιπόν, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει κανείς σε επαγγελματικό επίπεδο. Πολλές φορές έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πολιτιολόγοι και μετά καταλήγουν να είναι μπάρμεν στο Λονδίνο. Δεν σημαίνει αυτό τίποτα όμως. η παιδεία πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι αυτοσκοπός σε κάποιο βαθμό, ότι έχει την αξία της και δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι δύσκολο και το επάγγελμα του διδάσκοντος. Και μειώνεται ο αριθμό των ε, διδασκόντων και αυτών που θέλουν να ασχοληθούν με την παιδεία. Αυτό οδηγεί και σε μία, μία μείωση του επίπεδου παιδείας. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε πραγματισμό γιατί με αυτόν τον τρόπο μονάχα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ όλους που εργάστηκαν. Μεγάλη αξία έχει. Θα γίνει έξοχη δουλειά θα δοθεί προσανατολισμό, θα επαναπροωθηθεί μια στρατηγική που σίγουρα θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να αναδιατυπωθεί όσον αφορά κάποιε στοιχέ τη βάση κριτηρίων. Πού αναφέρατε. Λοιπόν, τι πληροφορίε να σα δώσω. Ο του εισηγητή θα υποβάλει το σχέδιο κειμένου στη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου της Επιτροπής μας, 17-18, η ψηφοφορία θα γίνει στις 19 Απριλίου. Καλώς. Πάμε σε σημαντική συνάντηση που έχουμε οργανώσει. Γνωρίζετε ότι σχετίζεται με την έκθεση. Ήταν χρήσιμο να έχουμε πληροφόρηση από την DG EAC και την ευχαριστώ που είναι εδώ για τη μελέτη που έγινε για το θέμα της παιδείας και της κατάρτισης και για θέματα καινούργια που έχουν αναδειθεί, που δεν είχαν θυγεί. Μόλις δημοσιεύτηκε αυτό το έγγραφο του ελέγχου αυτού, της εποπτείας αυτής, ευχαριστούμε την DGAC e για τα βασικά συμπεράσματα. Μας δόθηκαν δύο τόμοι. Ένας αφορά την υπερεθνική ανάλυση των διαφόρων θεμάτων και δεύτερον έχουμε κάθε χώρα από τις 28, τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα της κάθε χώρας. Είναι σημαντικό αυτό, διότι ε, θα είναι χρήσιμα κάποια στοιχεία που περιέχονται, χρήσιμα για την έκθεσή μας. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπείται εδώ γι' αυτό. Ευχαριστώ τον Μάικλ Τόιτς, επικεφαλής της μονάδας, και δεν Μάιερ, ε, μονάδας, υπεύθυνη για θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ευκαιρία να παρουσιάσω την έκθεση αυτή. Να σας πω εν συντομία περί τίνος πρόκειται. Και οι συναδελφοί μου θα παρουσιάσουν και άλλα στοιχεία από τα πορίσματά μας για την ευρωπαϊκή παιδεία. Βλέπετε τώρα τις ε, διαφάνειες και εκεί μπορείτε να έχετε μια πλήρες εικόνα. Εδώ το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι ο στόχος μας δεν είναι να περιγράψουμε το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά να κάνουμε μια ανάλυση των προβλημάτων, να χρησιμοποιήσουμε τα ποσοτικά στοιχεία που έχουμε για να εντοπίσουμε αφενός τα προβλήματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν και από την άλλη πλευρά να δούμε ποιες είναι οι πολιτικές ε, τάσεις και εξελίξεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδυάζοντας αυτά τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία μπορούμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι πιο σημαντικές πολιτικές προκλήσεις στο, στον τομέα της παιδείας. Θέλουμε να δούμε λοιπόν και πού βρίσκονται τα προβλήματα αλλά και πού βρίσκονται οι βέλτιστες πρακτικές στα κράτη-μέλη. Άρα η έκθεση αυτή είναι μια έκθεση η οποία θέλει να αντιμετωπίσει ε, οριζόντιες προκλήσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα. Από την άλλη μεριά έχουμε 28 σύντομες εκθέσεις ανά κράτος μέλος που παρουσιάζουν τις πιο σημαντικές προκλήσεις, τα πιο σημαντικά προβλήματα για κάθε συγκεκριμένο κράτος μέλος και τις αντίστοιχες πολιτικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα σε κάθε χώρα. Γιατί το κάνουμε αυτό. θέλουμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική για την παιδεία που να βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία για να μπορούμε να δούμε κατά πόσο μπορούν να είναι έφορε οι νέε πρωτοβουλίες για τη σχολική πολιτική τουλάχιστον να βασίζονται σε μια πραγματική τεκμηρίωση και θέλουμε να συνεργαστούμε και με τα κράτη-μέλη για την καλύτερη μεταλαμβάνευση των βελτίστων πρακτικών γιατί αυτό, αυτή η ανταλλαγή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για να υποστηρίξει ακόμα περισσότερο τι προσπάθειε των κρατών μελών. Αν βλέπει κανεί ότι ένα άλλο κράτο μέλο κάνει τα πράγματα καλύτερα, προφανώ αυτό μπορεί να βοηθήσει την πρόοδο. Αυτά λοιπόν υπό μορφή τη εισαγωγή και η συνάδελφό μου τώρα θα περάσει στα πιο επιμέρους συγκεκριμένα θέματα που είναι οι προκλήσει σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθώ. Α, δεν δουλεύει το σύστημα. Α, δουλεύει. δουλεύει. Λίνα Μάιερ είναι το όνομά μου. Αν σας ενδιαφέρει αυτό που δημοσιεύσαμε, εκεί στο τραπέζι, στην είσοδο της αίθουσας, έχετε το έντυπο και διάφορα φυλάδια, ε, πάρτε ό,τι θέλετε και έχουμε και κάποιες από τις εκθέσεις κατά χώρα εκεί. Είναι η τέταρτη έκδοση της εκθέσεως που διαιρείται σε τρία τμήματα. Το πρώτο δείχνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την παιδεία και την κατάρτιση. Μετά έχουμε ένα τμήμα που παρουσιάζει ποσοτικός πώς την κατάσταση, τι δείχνει το σύστημα βαθμολόγησης και έχουμε τρίτο τμήμα. Δείχνει το τι μπορούμε να πετύχουμε όσον αφορά διάφορες δράσεις, διαμόρφωση πολιτικής κλπ. Μία έκφραση που χρησιμοποιούμε στο πρώτο τμήμα είναι ένας όρος. Πασίγνωστος στους πανεπιστημιακούς κύκλους. Λιγότερο στο χώρο της πολιτικής. Μιλάμε για εκπαιδευτική φτώχεια. Και τι κινδύνους δημιουργεί. Τι εννοούμε με αυτή την εκπαιδευτική παινία. Στο δημοσίευμα εκεί που βλέπετε ε, αυτό είναι ένα έντυπο που είναι προϊόν του ερευνητικού προγράμματος. Δείχνει τι στοιχεία υπάρχουν όσον αφορά αυτή την εκπαιδευτική παιδεία, παινία. Συγγνώμη. Στο έντυπό μας αναφερόμαστε στην έλλειψη βασικών δεξιοτήτων. Βλέπετε εδώ κάποια αποτελέσματα την έρευνα του ΟΣΑ. Μεγάλο ποσοστό των φοιτητών όταν είναι 15 των σπουδαστών δεν κατέχουν τις βασικές δεξιότητες. Έχοντας πάει στο σχολείο για πάνω από 10 χρόνια. Πολλοί από αυτούς όμως τους μαθητές έχουν πολύ ανεπαρκείς δεξιότητες όσον αφορά την ανάγνωση, τα μαθηματικά κλπ. Αυτό είναι ενισχυτικό. Βλέπετε στο διάγραμμα. Έχουμε σύστημα βαθμολόγηση και γι' αυτό. Μέχρι το 2020 χρησιμοποιούμε αυτό το σύστημα. Μειώνουμε το ποσοστό αφαιρούμε το ποσοστό αυτό των μαθητών που δεν έχουν επαρκείς δεξιότητες στο 15%. Στα μαθηματικά είμαστε στα 22% περίπου. Βλέποντας τώρα τους μαθητές και το κοινωνικό και οικονομικό τους υπόβαθρο, κατάσταση γονέων, οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού στο οποίο ανήκουν, του σπιτιού τους, βλέπουμε ότι είναι διασκορπισμένα τα στοιχεία, ευρύ το φάσμα. Μεγάλη διαφορά εκείνων που αριστεύουν σε σύγκριση με εκείνους που δεν τα καταφέρνουν. Τα παιδιά από τα πιο χαμηλά επίπεδα είναι στο 36%. 36% από τα παιδιά που είναι από χαμηλά στρώματα οικονομικά δεν τα καταφέρνουν. Σε κάποια κράτη-μέλη είναι διαφορετική κατάσταση. μέχρι 50% των νέων παιδιών, μέχρι 15, δεν κατέχουν τις βασικές ε, γνώσεις σε κάποια κράτη-μέλη. Ποια είναι τα συμπεράσματά μας. Αυτή η εκπαιδευτική φτώχεια, η έλλειψη των βασικών γνώσεων, κινείται σε πολύ ψηλά επίπεδα και υπάρχει δυσανάλογη διάδοση στην κοινωνία μας, στις κοινωνίες μας και στις κοινωνικο-οικονομικές ομάδες. Βλέποντας τα στοιχεία για τις δαπάνες, βλέπουμε ανησυχητικές τάσεις. Τα κράτη-μέλη κάνουν περικοπές όσον αφορά την παιδεία. Αυτό δεν σχετίζεται με τη δημογραφική εξέλιξη όσον αφορά τους μαθητές. Βλέπετε εδώ το γράφημα, τη γραφική, γραφική παράσταση. Δύσληπτη η παρουσίαση αυτή των στοιχείων. Έχουμε τέσσερα τεταρτημόρια και εκεί μοιράζουμε τα στοιχεία. Τι λέει όμως η γραφική παράσταση έχουμε αλλαγή όσον αφορά τους πληθυσμούς των μαθητών. Σε σχέση με τον οριζόντιο και τον κάθετο άξονα. Στον οριζόντιο άξονα έχουμε πρόσφατες εξελίξεις. Στον κάθετο άξονα έχουμε μελλοντικέ εξελίξεις. Και έχουμε τις κουκίδες. Οι πορτοκαλί κουκίδες δείχνουν τις αυξήσεις. Όταν έχει αύξηση του ε, προπολογισμού στα κατημέλη και στα, με το πορφυρούν χρώμα έχουμε τις μειώσεις. Στο τέταρτο τετατημόριο έχουμε τις περικοπές βλέπετε. Έχουν γίνει περικοπές εκεί, αλλά έχουν και φοιτητικό πληθυσμό που αυξάνεται. Ο συνδυασμός των δύο δεν είναι καθόλου καλός. Μπορεί κανείς να πει ότι ίσως να έχουμε βελτιώσεις απόδοση στην παιδεία. Δύσκολο να το διαπιστώσουμε αυτό. Να εντοπίσουμε την απόδοση στον τομέα της παιδείας. Εμείς βλέπουμε περικοπές στις χώρες. Καθόλου ενθαρρυντικό. Και ξανά διαγράμμα. Τα παιδιά που φεύγουν νωρίς από το σχολείο δείκτες ε, του πλαισίου Ευρώπη 2020. A, B, C, D τα τεταρτημόρια. Κάποιες χώρες κάνουν περικοπές. Μάλλον κάποιες χώρες τα πηγαίνουν καλά, κάποιες λιγότερο καλά. Ανησυχούμε για εκείνους που ανήκουν στο τέταρτο τεταρτημόριο, το D, πάνω δεξιά στην οθόνη. Εμείς θέλουμε μόνο 10% των παιδιών να φεύγουν προώρα το σχολείο. Οι χώρες στο τετατημόριο D έχουν υψηλότερο επίπεδο. Πάνω από 10%. Και δεν έχουμε και καμία πρόοδο σε αυτές τις χώρες. Λοιπόν, στην έκθεση τι κάνουμε. Μπαίνουμε στις λεπτομέρειες. Ποιοι είναι αυτοί οι μαθητές που φεύγουν προώρα από το σχολείο. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο φίλων. Τα κορίτσια τα πηγαίνουν πολύ καλύτερα τα αγόρια. Όταν γεννιέται κανείς σε μια χώρα που στη, όταν μένει στη χώρα που γεννήθηκε κάποιος ε, μάλλον ή σε χώρα της αλλοδαπής υπάρχει διαφορά. Αυτοί που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και ζουν σε άλλη χώρα, ε, είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που φεύγουν, που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, σε σχέση με αυτούς που έχουν μείνει στη χώρα τους. Λοιπόν, εξαρτάται το ποσοστό εκείνων που έχουν φύγει πρόωρα, εξαρτάται πότε έφτασε το παιδί στη χώρα διαμονής και πότε ξεκίνησε να πήγαινε στο σχολείο, σε αυτή τη χώρα. κοιτάμε τα άτομα που είναι 18 μέχρι 24 ετών που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση. Εκείνοι που φεύγουν πριν την υποχρεωτική εκπαίδευση μπαίνουν στα υψηλά ποσοστά αποχωρούντων. Αν μείνουν περισσότερο στη χώρα έχουν άλλα ποσοστά σε σχέση, πιο ψηλά ποσοστά σε σχέση με τον τόπιο πληθυσμό. Αυτό δείχνει ότι όταν θέλουμε να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε την ε, προ, πρόορη σχολική εγκατάλειψη ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Τώρα, εδώ θέλω απλώς να δείξω κάποια πράγματα τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πιο ποιοτική εκπαίδευση και να δούμε τι λένε τα δεδομένα, τι δείχνουν τα ερευνητικά πορίσματα. Ένα από αυτά είναι το θέμα της περιεκτικότητος. Και εδώ μιλάμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της διδασκαλίας. Ξέρουμε ότι οι διδασκόντες είναι πάρα πολύ σημαντικοί για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα που παίρνουμε από τη σχολική εκπαίδευση και η έρευνα του ΟΣΑ Και η έρευνα αυτή δείχνει ότι οι διδάσκοντες δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν την πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου και χρειάζονται περισσότερη παιδεία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ε, πολιτιστική διαφορετικότητα και τις διαφορετικές ανάγκες που έχουν ε, οι μαθητές και τους μαθητές με ειδικέ ανάγκες. Σύγχρονως υπάρχουν ανάγκες πιο εξειδικευμένων στρατηγικών για να αντιμετωπίσουμε στην ανώτερη παιδεία που έρχονται με ειδικέ ανάγκες ώστε να μπορέσουν και στο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό επίπεδο να προσαρμοστούν. Αυτά λοιπόν είναι κάποια αποτελέσματα. Και ο Μάικελ θα σας πει κάτι περισσότερο για τα παραδείγματα αναχώρα. Ευχαριστώ λέει ο Μάικελ. Έρχεται εδώ πέρα κάποια α, παραδείγματα. Το monitor βέβαια έχει συγγραφεί στα αγγλικά. Έχουμε όμως μερικά σημαντικά α, μηνύματα και για κάθε γλώσσα φυσικά αντιμετωπίζουμε μαζί κάπως τις χώρες που μιλάνε αυτές τις χώρες. Και παραδείγματος στην Ιταλία μιλάμε για τα Ιταλικά αλλά και για τα Αγγλικά, στην Ουγγαρία για τα Ουγγρικά αλλά και τα Αγγλικά. Έχουμε τις πιο σημαντικές γλώσσες στην παιδεία για κάθε χώρα. Η αναλύση, λοιπόν για την εγκατάλειψη του σχολείου θα πρέπει να τα εξετάσουμε λίγο πιο προσεκτικά και βλέπουμε τώρα το, το θέμα της συμπερίληψης. Έχουμε κάποιες μελέτες που έχουν γίνει για το τι κάνει η Σουηδία για να αντιμετωπίσει τα παιδιά που είναι παιδιά μεταναστών ή μετανάστες που έρχονται. Η Σουηδία έχει ήδη εδώ και πολλά χρόνια ξεκινήσει μια μεγάλη για να έχει μια, μια έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων, διαγνωστικές μελέτες ή επίσης να υπάρξει ιδιαίτερη εκπαίδευση των ε, καθηγητών για τα θέματα αυτά, εισαγωγικά μαθήματα και κτλ. Λοιπόν, τώρα δεν, ε, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τα σουηδικά ή όχι. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το παράδειγμα της Ιταλίας στον τομέα της ε, ποιότητας. Έχουμε κοιτάξει πιο προσεκτικά την τωρινή μεταρρυθμίση που λαμβάνει η χώρα στην Ιταλία και ξέρει και η πρόεδρος ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα που έχει παίξει κάποιο ρόλο σημαντικό και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που το έχει προωθήσει Ο στόχος είναι να υπάρξει μεγαλύτερη αυτονομία του σχολείου, καλύτερη αξιολόγηση των διδασκόντων και μια διαδικασία μάθησης η οποία βασίζεται περισσότερο στην πρακτική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το λεγόμενο ψηφιακό πανεπιστήμιο στη Γαλλία, η οποία έχει αγωνιστεί ιδιαίτερα να μπορέσει να αναπτύξει μια καλύτερη εθνική στρατηγική σε ό,τι αφορά την ψηφιακή μάθηση στο πανεπιστήμιο. Δίνουμε λοιπόν τέτοια παραδείγματα γιατί νομίζουμε ότι τα παραδείγματα αυτά είναι σημαντικά και μπορούν να είναι σχετικά και με τις ανάγκες άλλων κρατών μελών όταν θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε μια μεταρρύθμιση. Παραδείγματο χάρη, η τσεχική δημοκρατία, η Σλοβακία μπορούν να υποφεληθούν από τις εμπειρίες που έχουν άλλες χώρες όπως η Ιταλία στον τομέα της μεταρρύθμισης και η ελπίδα μου είναι ότι και για σας θα είναι ενδιαφέρουσα η ανατύπηση αυτής της έκθεσης και των παραδειγμάτων που δείχνουμε σε ποιους ακριβώς τομείς αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται πρωτοβουλίες μεταρρύθμισης στην Ευρώπη. Αυτά είναι λοιπόν ένα, μια πρόγευση, αν θέλετε, ένα απεριτήφ για την πλήρη έκθεση που θα έχετε στη διάθεσή σας εν καιρό. Σας ευχαριστώ, Λεγική Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη ενημέρωση που μας κάνατε και για τις ενδιαφέρουσες ε, θέσεις και ενδιαφέροντα θέματα που παρουσιάσατε. Αυτό το monitor λοιπόν, αυτή η έκθεση που εκπονήσατε είναι μεγάλο ενδιαφέροντος διότι όπως γνωρίζετε πολύ καλά στην έκθεσή μας ασχολούμαστε με το θέμα της εκπαίδευσης εν ώψη του 2020, τον στόχο 2020 και είναι σημαντικό λοιπόν στην προσπάθειά μας να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις προκλήσεις, πραγματικές προκλήσεις και κάποιες ε, προσεγγίσεις ε, πρέπει να διαρευνηθούν. Αυτό απαιτείται ιδιαίτερα στις προσπάθειες που κάνουμε. Μεταξύ άλλων το θέμα της, της εκπαιδευτικής φτώχειας και του κινδύνου των κοινωνικών διαφοροποίησεων, της αυξήσεως του κοινωνικού χάσματος των φατήμπρων στο σχολείο είναι πολύ σημαντικό. Και τα άλλα θέματα. Η ποιότητα της μάθησης είναι θέματα αυτά που τα συζητήσαμε και πριν. Αναφερθήκατε βέβαια όταν συζητούσαμε πριν την έκθεση του συναδέλφου Κρασνοντέψκη τα θύσαμε αυτά. Η Πέτρα έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και την Κομισιόν για την παρουσίαση αυτής της τόσο ενδιαφέρουσα ε, μελέτης. Έχω να κάνω τώρα ένα συμπληρωματικό ερώτημα προς εσάς. Δίνεται καταρχήν ένα πίνακα όπου αναφέρεται το ποσοστό απασχόλησης ανεξάρτητα από το επίπεδο παιδείας. Και καταλήγεται στο συμπέρασμα, μάλλον σε συνάντηση με την ε, σχολική εκπαίδευση, <coughs> ότι για, την, ε, ε, για το μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης έχετε ένα ποσοστό το οποίο διστάζεται κατά 100. Σκέφτομαι τώρα άλλες χώρες όπως είναι η Γερμανία ή όπως είναι η Αυστρία όπου υπάρχει ένα πιο πολύπλοκο σύστημα το οποίο για τα μεσαία εκπαιδευτικά επίπεδα συνδυάζει την εργασία και την εκπαίδευση. Μπορείτε να δείτε αν είναι καλύτερα τα αποτελέσματα σε χώρες όπως αυτές οι οποίες έχουν ένα σύστημα πρακτικής ε, εξάσκησης και αν είναι καλύτερα τα πράγματα στις χώρες αυτές σε σχέση με άλλες χώρες όπου είναι μονάχα στο σχολικό επίπεδο η εκπαίδευση και δεν υπάρχει τόσο στενή σύνδεση με τις επιχειρήσεις. Εμείς στη Γερμανία και φαντάζομαι και στην Αυστρία θεωρούμε πάντα ότι το σύστημά μας είναι τόσο καλό που θα έπρεπε όλες οι χώρες της Ευρώπης να το υιοθετήσουν και πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο διτό σύστημα παιδείας μπορεί να εξασφαλίσει ότι υπάρχει μεγαλύτερη απασχολησιμότητα των νέων που δεν έχουν τόσο υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα. Αλλά ακριβώς επειδή η εκπαίδευση αυτή βρίσκεται πιο κοντά στο χώρο εργασίας μπορεί να προσφέρει περισσότερο. Έτσι το λέμε εμείς και εμάς μας φαίνεται προφανές. Αλλά ξέρω ότι υπάρχουν και άλλες ε, απόψεις. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο και οι στατιστικές καταδεικνύουν αυτό ότι ακόμα και άνθρωποι με περιορισμένα εκπαιδευτικά προσόντα μπορούν χάρη σε αυτό το σύστημα να έχουν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης από ό,τι σε άλλα συστήματα. Ευχαριστώ κύριος Καστοντέσκη. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρον υλικό. Θα τα συμπεριλάβουμε αυτά, τις προτάσεις αυτές που ακούσαμε στη δική μας έκθεση. Δύο ερωτήσεις έχω. Η μία αφορά τις μεγάλες διαφορές μεταξύ κάποιων χωρών ας πούμε πολύ κακές επιδόσεις στα μαθηματικά. Βλέποντας τη χώρα μου, την Πολωνία, πάντα έχει καλές επιδόσεις. Μια χώρα που είναι κοντινή μας πολιτισμικά και ιστορικά, η Ουγγαρία τα πάει χάλια. Και υπάρχουν και οικονομικές εξελίξεις. Φαντάζομαι ποια είναι τα αίτια των διαφορών και τι συμβαίνει στη Βουλγαρία. Ποιοι είναι οι λόγοι των διαφορών. Είναι μόνο τα εκπαιδευτικά συστήματα για τις κακές επιδόσεις ή συμβαίνει κάτι άλλο. Δεύτερον, η διαφορά μεταξύ των φύλων. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή. Όταν μιλάμε για τις έμφυλες διαφορές μιλάμε για την κακή θέση των γυναικών, προβλήματα που έχουν οι γυναίκες για πρόσβαση στην αγορά. Στην παιδεία όμως έχουμε άλλο πρόβλημα. Δεν τα πηγαίνουν καλά τα αγόρια, οι άντρες, στις επιδόσεις. Σε κάθε επίπεδο και σε πανεπιστημιακό επίπεδο, αν δείτε τις λεπτομέρειες, σε γνωστά πανεπιστήμια, τα κορίτσια τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα τα αγόρια. Και υπάρχουν σχετικά στοιχεία που το δείχνουν αυτό. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ χωρών επίσης. Σε κάποιες χώρες διαφορές κοριτσιών αγοριών δεν είναι τόσο μεγάλες όπως τη Βουλγαρία και αλλού. Πώς το εξηγείτε αυτό. Οφείλεται η διαφορά μόνο σε οργανωτικά θέματα της παιδείας ή κάτι άλλο. Φταίει οικονομική κατάσταση. Δεν ξέρω. Άλλος, πολύ σύντομα, από ό,τι άκουσα, είδα τι συμπεριλαμβάνεται, τι συμπεριλαμβάνεται. Δύσκολε συγκρίσει. Εκεί που έχουμε τι μεγάλε επιχειρήσει και εκεί που έχουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, άμα κάνουμε τι συγκρίσει εκεί, έχουμε άλλε αφετηρίε. Το διτό σύστημα, το αυστριακό και το γερμανικό είναι πολύ διαφορετικό από το ιταλικό. Και έχει σημασία αυτό. Χρειάζεται μηχανισμό που λαμβάνει υπόψη αντικειμενικά στοιχεία για τι χώρε. Ερώτηση. Κάνατε αναλύσεις. Γίνεται παραλληλισμός μεταξύ επίπεδου καταρτήσεως που εξασφαλίζεται μέσω των σχολικών προγραμμάτων ή επαγγελματική κατάρτισης με τον, ε, την έλλειψη δεξιοτήτων σε σχέση με τις ανάγκες των θέσεων απασχόλησης. Μπορεί να διευκρινιστεί αυτό. Ανάλογα με τα επίπεδα υπάρχουν και δυνατότητε απασχόλησης. Γύηση γι' αυτό βέβαια. Δεν υπάρχει βεβαιότητα όσον αφορά την αντιστοιχία σπουδών και εργασίας. Όμω, όσο πιο χαμηλό το επίπεδο τη εκπαίδευση, τόσο περισσότερε πιθανότητε η απασχόληση να είναι ε, σε χαμηλότερα επίπεδα, με χαμηλότερε απαιτήσει. Όταν κάποιος σπουδάζει, σταματά και πάει στη δουλειά μετά κατευθείαν. Τι προβλήματα δημιουργούνται. Το μελετήσατε. Ίσως είναι κάτι που θα έπρεπε να αναλυθεί. Ο κύριος Μαραγάλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μερικές σύντομες σκέψεις. Πρώτα απ' όλα, Εγώ είμαι για την ποιότητα της έκθεσης και των στατιστικών στοιχείων που έχουν παρουσιάσει. Είναι συναρπαστικά αυτά. Παρά το γεγονός ότι είναι κυρίως στατιστικού χαρακτήρα η έκθεση, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στις ε, ευρωπαϊκές στατιστικές, αλλά δεν ξέρω για, για τις εθνικές στατιστικές αν είναι αξιόπιστες ή εξάλλου αν είναι πραγματικά συγκρίσιμες μεταξύ τους, αν έχουμε τα ίδια κριτήρια που χρησιμοποιούμε. Θα ήθελα να εξασφαλιστεί αυτό δεύτερον. Για την σχολική εγκατάλειψη, την πρόορη σχολική εγκατάλειψη. Εγώ παρακολουθώ αυτό το οποίο γίνεται στην χώρα μου, στην Ισπανία, συγκεκριμένα στην Καταλωνία σύμφωνα με τη μελέτη, για μένα θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να έχουμε δείκτες για την εξέλιξη ε, των οικονομικών δικτών και της σύνολης οικονομίας μιας χώρας. Στην ε, χώρα μας, στην εποχή της οικονομικής ε, άνθησης, στην οικονομικό τομέα και στον τουρισμό, αυτό αύξησε άμεσα και μαζικά την σχολική εγκατάλειψη, γιατί πάρα πολλά παιδιά φεύγανε από το σχολείο, τους πέραν από το χέρι οι εργοδότες, τους δίνανε αμέσως δουλειά και έλεστα Ακόμα και αν ήταν προσωρινή εργασία και επισφαλής. Τα επόμενα χρόνια αυτό το οποίο αντιστάθμισε τα πράγματα ήταν η εγκατάλειψη των μεταναστών, εγκατάλειψη της, του σχολείου από τους μετανάστες που γυρίσαν στις χώρες τους λόγω της οικονομικής κρίσης. Θέλω να πω ότι υπάρχουν διαφορετικοί ε, παράγοντες που επηρεάζουν το παραγωγικό και το εκπαιδευτικό σύστημα παράλληλα. Όπως είπε λοιπόν και ο κύριος Μοργάνο, είναι πολύ πιο δύσκολο να υπάρξει σύγκριση όταν εμείς κοιτάμε τα θέματα της εργασίας και της ε, εκπαίδευσης κάτι το οποίο μπορεί να είναι ναι. κατάλληλο μοντέλο για την Αυστρία και τη Γερμανία, ενδεχομένως μπορεί να μην είναι το καταλληλότερο για οικονομίες όπως είναι η Ισπανική οικονομία. Γι' αυτό νομίζω θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να βρείτε έναν τρόπο να καταδείξετε καλύτερα τους μηχανισμούς αυτούς μεταξύ εργασίας και εκπαίδευσης που να είναι προσαρμοσμένοι στις διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Κάτι άλλο, μια γενικότερη παρατήρηση που δεν έχει καμιά σχέση με την έκθεση αυτή. Είπα προηγουμένως, μιλώντας για την έκθεση του κ. Κασνοβιέσχη, ότι έχουμε ε, το σύστημα της Μπολόνιας και την, ε, τον έρασμο, αλλά όχι στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια παιδεία. Έχουμε μονάχα το σύστημα πίσα για την ε, παιδεία. Αλλά αυτό είναι ένα παγκόσμιο σύστημα. Εγώ σκασίλαμε τι γίνεται στην Νότια Κορέα ή στην ε, Σιγκαπούρη. Θα με ενδιαφέρει περισσότερο να μπορώ να συγκρίνω την ε, Ισπανία και την Πορτογαλία με τη Βουλγαρία ή τη Σουηδία. Θέλουμε να έχουμε τέτοια εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν τα έχουμε. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας χώρος εργασίας που μπορεί να είναι πολύ σημαντικός και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικός για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, Ευχαριστώ. Και εγώ έχω δύο ερωτήσεις εντάχει. Η πρώτη. Λέτε σε κάποια φάση ότι ο θεμελιώδες είναι να δούμε και τι γίνεται στην τοβάθμια εκπαίδευση. 25% των πτυχιούχων εργάζονται σε θέσεις που, ε, στις οποίες εργάζονται περισσότερο από εκείνους που δεν έχουν τρίτο βάθμιο πτυχίο που δεν απαιτούν σε θέση, δεν απαιτούν πτυχίο απαραίτητα. Και δεν υπάρχει τέριασμα μεταξύ δεξιοτήτων και θέσης απασχόλησης. Καλό λοιπόν, εάν να μπορέσετε να μας αναλύσετε περισσότερα τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι πιο ικανά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις με την αγορά εργασίας να υπάρχει καλύτερη αντιστοιχεία γνώσεων με αγορά εργασία. Αναλύοντα τα στοιχεία, όσον αφορά του πτυχιούχου, τα ξέρω αυτά. Η Ιταλία έχει μικρότερο ποσοστό πτυχιούχων σε σχέση με, με άλλες χώρες. Και δεν υπάρχει τόσο πολύ καλή αντιστοιχεία μεταξύ ε, πτυχιούχων και θέσεων εργασία. Έχουμε λήψεις και κενά σε εκείνους που καταλείπουν νωρί την εκπαίδευση, τους early leavers. Σωστό αυτό που είπατε, σημαντικό. Υπάρχει διπλή παινία, εκπαιδευτική τη αυτή, αλλά και αυξανόμενη κοινωνική διαφοροποίηση όσον αφορά την πρόσβαση και στη συνέχιση των σπουδών. Διπλό divide που αντιμετωπίζουμε. Είναι ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κ. Κρασνοντεύσκη ότι τα κορίτσια δεν εγκαταλείπουν τόσα πολλά ε, το σχολείο και έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή όσον αφορά την ανώτερη εκπαίδευση και τους τυχιούχους. Μήπως υπάρχει θέμα προσανατολισμού. Ίσως είναι διευθυντικό το πρόβλημα και δεν αφορά κάποιο μονομένο σύστημα, αλλά μια διάθεση που έχουν τα κορίτσια να προσπαθούν περισσότερο. Διότι ξέρουν ότι από αυτό εξαρτάται και το μέλλον της δουλειάς τους. Πιστεύετε ότι είναι κάτι που έχει σχέση με διαφορετικά στοιχεία ή όχι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το ερώτημά σας. Αν μπορώ να απαντήσω λίγο εν συντομία, επανέρχομαι σε αυτά που είπε η κυρία Κάμερβετ για τα διτά συστήματα όπως ε, στην ε, Αυστρία και τη Γερμανία που λένε γενικά ότι όσο πιο υψηλή οι όσο πιο ψηλή είναι η εκπαίδευση, τόσο μεγαλύτερη η συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Δηλαδή χώρες που έχουν πιο ψηλή τριτογενή εκπαίδευση τα καταφέρουν πολύ καλύτερα. Αυτό που λέτε εσείς είναι, το πλεονέκτημα είναι ότι δεν είναι τόσο μεγάλη η απόσταση ανάμεσα στο χώρο εργασίας και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στη Γερμανία και την Αυστρία, αλλά και στις κάτω χώρες όπου άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαμηλή γενικά παιδεία μπορούν να έχουν καλές ευκαιρίες ε, πρόσβασης στην αγορά εργασίας. φυσικά ε, επηρεάζεται η πρόσβαση στην αγορά και από την μορφή της ε, οικονομικής δραστηριότητας. Εμείς έχουμε κάνει μονάχα μια επισκόψη για τα τελευταία 20 χρόνια. Εκεί που δεν μπορούμε λοιπόν να ξέρουμε συνολικά τι γίνεται, αυτό το οποίο ε, δεν είμαι τόσο σίγουρος είναι για τον ενδιάμεσο αυτό επίπεδο Ακόμα και στη Γερμανία και στην Αυστρία λόγω του διτού συστήματος υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκπαιδευτική παινία όπως λέγεται και έχουν για αυτό το λόγο δυσκολία απασχόλησης. Αυτό που είπε ο κ. Καρνοντεύσκη για τη σύγκριση Πολωνίας και Ουγγαρίας. Η Πολωνία έκανε μια μεγάλη μεταρρύθμιση πρόσφατα και με τον τρόπο αυτό έχει κάπως διαφοροποιηθεί από την Ουγγαρία όπου παίζει μεγαλύτερο ρόλο η συμμετοχή, ο ρόλος των γονέων και του οικονομικού συστήματος. Η Πολωνία λοιπόν έχει καταφέρει πολύ καλά τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις κλασικές δεξιότητες, γραφή και ανάγνωση. και έχει γίνει και αρκετή πρόοδος χάρη στη μεταρρύθμιση σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των δασκόντων. Τώρα, για τη διαφορά μεταξύ των φύλων, όπως είπε και η πρόοδος, έχουν μεγαλύτερα προβλήματα τα αγόρια από τα κορίτσια. Δεν φαίνεται να υπάρχει μια μεγάλη τροποποίηση αυτού του σύστηματος και αυτό φαίνεται ότι δεν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το ένα άλλο πράγμα που δεν έχει να κάνει με το εκπαιδευτικό σύστημα είναι η διαφορά ανδρών και γυναικών σε ό,τι αφορά το χώρο εργασίας. Πρέπει όμως να αντιμετωπίσουμε περισσότερο την διάσταση του φύλου στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ε, σας λέω πάλι ότι σε σχολικό επίπεδο τα αγόρια έχουν τα περισσότερα προβλήματα, αλλά αντίστοιχα στο χώρο εργασίας είναι οι γυναίκες. Ο κύριος Μοργκάνο λοιπόν επίσης, ε, αν κατάλαβα καλά. Αναφέρθηκε στο θέμα της περαιτέρω κατάρτισης που μπορεί να έχει κάποιος όταν έρχεται στην αγορά εργασίας και ο κύριος Μαραγκάλ αναφέρθηκε στο θέμα της Ισπανίας όπου υπήρξαν σημαντικά προβλήματα στην αγορά εργασία, κυρίως στον οικοδομικό, τον κατασκευαστικό κλάδο και όπου προσελκύστηκαν πάρα πολλοί νέοι να αποχωρήσουν από το σχολείο για να περάσουν στο χώρο εργασίας και αυτή τη στιγμή βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι άνεργοι και έχουν τεράστια προβλήματα. Και οι συζητήσεις που κάναμε έδειξαν και η Ισπανία προσπαθεί να αναπτύξει νέα υποδείγματα εκπαίδευσης γιατί όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει δεν ήταν ιδιαίτερα βιώσιμα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Επίσης, όπως είπε ο κύριος ε, Μαραγκάλ, εμείς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα του ΟΣΑ, τις στατιστικές του ΟΣΑ. Εκεί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδόν όλα συμμετέχουν. Χρησιμοποιούμε επίσης τις δημοσίευσεις πέραν από το ΟΣΑ και τη, του, της Eurostat και αν έχουμε και άλλες εθνικές στατιστικές θα χρησιμοποιούμε αυτά. Φυσικά οι στατιστικές μας προέρχονται κυρίως από το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Αυτά που είπε η κυρία Κώστα, η για την ε, αναντιστοιχία στο πανεπιστημιακό επίπεδο, είδαμε να έχει αυξηθεί αυτό το ποσοστό. Υπήρξε στο παρελθόν κάποιο πρόβλημα με την ποσότητα. Υπήρχαν χώρες που είχαν πολύ χαμηλό επίπεδο τριτογενούς εκπαίδευσης, αλλά βλέπουμε τώρα σε όλη την Ευρώπη να έχει αυξηθεί και το ποσοστό της αποχώρησης από τον τρίτο βαθμίο ε, τομέα. εντάξει. Δεν νομίζω ότι θέλω να συμπληρώσω τίποτα σημαντικό σε αυτά που είπε ο Μιχάλης. Ανάλογα με το αν κανείς έχει κάποιο προσανατολισμό προσπαθούμε να δούμε αν παίζει ρόλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Ξέρουμε ότι είναι πολύ ψηλότερη η ρυθμή απασχολησιμότητας όταν κανείς έχει υψηλή εκπαίδευση, αλλά τελευταία παρατηρήσαμε ότι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν έχει αυξηθεί η απασχολησιμότητα, ενώ για τη δευτεροβάθμια ναι. Βέβαια είναι σίγουρο ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση αν δεν καταλήγει σε απασχόληση πολλές φορές φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας αυτό το είπε και ο Ισπανός σας συνάδελφος γενικά αυτοί που φεύγουν γρήγορα από το σχολικό σύστημα 60% από αυτούς είναι είτε άνεργοι είτε ανενεργοί και το υπόλοιπο 40% απασχολούνται. Είναι σοβαρό θέμα και βέβαια θέλουμε ο κόσμος να μένει στο εκπαιδευτικό σύστημα, να εκπαιδεύεται καλύτερα για να απασχοληθεί στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ δουλέψει στο Eurostat πολλά χρόνια και έχουμε εξετάσει πολύ καλά τα στοιχεία κατευθείαν από τις πηγές τον ΟΣΑ, από το Γιώργο και τα λοιπά και με το Γιουρίντιση η Βρυδίκη για να δούμε κατά πόσον είναι αξιόπιστα τα στοιχεία ή όχι ως προς τα διαφορετικά στοιχεία από διαφορετικές χώρες αν είναι συγκρίσιμα ευχαριστούμε Thank you so much. Grazie davvero. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την συνεισφορά σας πολυτιμότατη. πολυτιμότατη. Συμφωνώ ότι χρειάζεται να έχουμε συστήματα πιο ποιοτικά και σωστά στοιχεία όμως και δεδομένα. Ευχαριστώ. Μπορεί να είναι χρησιμότατη η συνεισφορά σας για την έκθεσή μας. Βασιζόμαστε στην εργασία μαζί σας. Mm. Και ευχαριστώ και τη μονάδα σας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το τμήμα της συζήτησης. Με τα χαράς καλωσορίζουμε. <laughs> Meeting. Allora, eh, το Γενικό Διευθυντή τη Γενική Διευθύνσεω Επικοινωνιών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Τίμο Πεσόνεν, ο οποίο είχε την καλοσύνη να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μα. Θα θυμόσαστε ότι όσον αφορά το σημαντικότατο θέμα της ενημέρωσης και την πολιτική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, εμείς ήμασταν Επιτροπή Αρμόδια στο Κοινοβούλιο βέβαια και θεωρήσαμε σημαντικό εν ώψη των θεμάτων θα αντιμετωπίσουμε να ενημερωθούμε όσον αφορά τη στρατηγική επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενημέρωση για τις πολιτικές που εφαρμόζει και τα σχέδια για την επικοινωνία σε συνεργασία με άλλους θεσμούς και κράτη-μέλη. Σε περίοδο κρίσεως που δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και πολιτισμική τίθεται θέμα της ποιότητας ενημέρωσης και στοιχείων που θα εμπεριέχει αυτή. Δεν είναι απλό το θέμα. Το εξετάσαμε ήδη. Όσον αφορά την ανάπτυξη της ευαισθησίας, όσον αφορά τα θέματα της ηθαγένειας, τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιες είναι οι αξίες, οι κοινέ που δημιουργούν ταυτότητα. Άρα χρειάζεται λεπτομερέστερη ενημέρωση και επικοινωνία μέσω των κοινωνικών μέσων. Νέα θέματα τίθενται. Νέα βάση χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως άλλαξαν και αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το θέμα. Έχουμε τώρα και το Euronews που μπαίνει στην αρμοδιότητα της DG Connect. Ενώ η Γενική Διεύθυνση για τον Πολιτισμό και την Παιδεία ακολουθεί άλλα προγράμματα. Έχει ιδιαιτερότητες η προσέγγιση με στη σφαιρικότητά της. Μας, ενδιαφέρεται πολύ, μας ενδιαφέρουν πολύ αυτά που θα μας πείτε. Θα υποβληθούν και ερωτήσει από συναδέλφου. Είναι πολύ στρατηγικό αυτό το θέμα και αυξάνεται η σημασία του η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα χρησιμοποιήσουν δουλειά που έχουν και τα κράτη-μέλη για την επικοινωνία στον αφορά το ΕΦΣΥ, για τι αδικέ επενδύσει και είναι κυκλική ενημέρωση. Χρειάζεται πρωτοβουλία και των κρατών μελών για το νέο Ταμείο Επενδύσεων. Θα συνεισφέρουν και βουλευτές στην προσπάθεια. Άρα χρειάζεται άλλο ύφο η επικοινωνία. Πολυσχηδή πρέπει να είναι η προσέγγιση. Με σφαιρική συμμετοχή. Σα ευχαριστώ για την παρουσία σας. Σας δίνω αμέσω το λόγο για ένα δεκάλεπτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που είμαι εδώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σα πω ότι μεγάλη τιμή είναι για μένα να είμαι εδώ και θέλω να σας υποστηρίξω για την υποστήριξή σα γιατί ακόμα και πριν από τη δική μου εποχή υπήρξε μεγάλη υποστήριξη από εσά στη διαδικασία του προπολογισμού. Εργαστήκαν τα δύο θεσμικά όργανα μαζί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί τα θέματα επικοινωνία είναι κυρίω αυτά τα οποία απασχολούν πάρα πολύ το Συμβούλιο. Και αυτό είναι πολύ σαφέ και εφέτος από τότε δηλαδή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Θα ήθελα τώρα να δω πιο ευραίος την συνεργασία μας και να σας πω τι προσπαθούμε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε την εισαγωγή των νέων προτεραιοτήτων επικοινωνίας της Κομισιόν και να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε καλύτερα και την συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων. έχετε αναφερθεί ήδη στις διαφορές της τρέχουσας επιτροπής από την προηγούμενη. Δεν είμαστε πια, δεν είμαστε πια υπεύθυνοι ούτε χρηματοδότες του Euronews, ούτε διαχειριζόμαστε το πρόγραμμα «Η Ευρώπη των πολιτών». Βέβαια η DigiConnect και άλλες γενικέ διευθύνσει ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Εμεί υπαγόμαστε άμεσα στον πρόεδρο Γιούγκερ μαζί με τη Γενική Γραμματεία του. Αυτό το οποίο θέλουμε να εστιάσουμε σε είναι οι 10 πολιτικές προτεραιότητες που έχει διατυπώσει η Κομισιόν. Και αυτό έχει γίνει δεκτό και από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι οι 10 πρωτοβουλίε του Πρόεδρου Γιούνκερ που παρουσιάστηκαν και σε εσά και στο Συμβούλιο. Σε αυτές εστιάζουμε κι εμείς. Και όπως είπε και η κυρία Πρόεδρε, Πρόεδρος, η πρωτοβουλία για την επένδυση στην Ευρώπη, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η οικονομική μεγέθυνση είναι η προτεραιότητα των προτεραιοτήτων. Όταν ακούτε συχνά ότι η Κομισιόν λέει ότι θέλουμε, θέλουμε να είμαστε μια πολιτική Επιτροπή. Αυτό δεν το λέμε μονάχα σε επίπεδο εκλογικό ότι ουσιαστικά έχει υπάρξει μια πολιτική διαδικασία που οδήγησε σε αυτή την Κομισιόν. Όχι, θέλουμε να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα υπέρ των πολιτών μας. Το μήνυμα λοιπόν του Προέδρου μας είναι ότι πρέπει να έρθουμε και πάλι σε επαφή με τους πολίτες μας, θα πρέπει να έχουμε καλύτερη επικοινωνία των σχεδίων και των στόχων της Κομισιόν και καλύτερη εστίαση στις προτεραιότητες. Έχουμε μεταρρυθμίσει την υπηρεσία του εκπροσώπου της Κομισιόν που υπάγεται στη δική μου γενική διεύθυνση. Οι εκπρόσωποι λοιπόν δεν είναι εκπρόσωποι κάθε γενικής διεύθυνσης αλλά είναι εκπρόσωποι του Προέδρου της Κομισιόν. Έχουμε λοιπόν ένα σχήμα το οποίο είναι λιγότερο πολυάριθμο και είναι και πιο αποτελεσματικός εκ τούτου επειδή και εγώ έχω λειτουργήσει ως εκπρόσωπος στο παρελθόν, νομίζω ότι λειτουργούμε πολύ καλύτερα τώρα. Όταν λέμε λοιπόν ότι θέλουμε να έχουμε καλύτερη επαφή με τους πολίτες, εσείς το ακούτε όταν είσαστε σε εκλογικές σας περιφέρειες, ότι θέλουν να ξέρουν περισσότερα για την Ευρώπη. Θα πρέπει κάθε μέρα να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας από πού προερχόμαστε, πώς ξεκίνησε το ευρωπαϊκό εγχείρημα, πώς δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα χρόνια και τους καιρούς. Και θα πρέπει να θυμηθούμε ποιες είναι οι βασικές μας αξίες, οι οποίες περιέχονται στις συνθήκες και στον, στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Εκεί εμπλέκεται η επικοινωνία. Πώς θα μπορέσουμε να τα μεταλαμβαδεύσουμε αυτά προς τους συμπολίτες μας. Αυτό που έκανε ο πρόεδρος Γιούκερ στην αρχή της θητείας του ήταν να ζητήσει από κάθε μέλος της Κομισιόν να πηγαίνει πιο συχνά στα κράτη-μέλη. Πηγαίνετε εκεί. Ελάτε σε επαφή με του πολίτες. Να είσαστε πιο ενεργός. Αυτό κάνει μια διαφορά. η επίτροποι είναι πιο συχνά παρόντες όχι μοναχά στις δικέ του χώρε, αλλά παντού στην Ευρώπη, σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε όλοι και να χρησιμοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες που μας δίνονται ώστε οι επίτροποι να έρχονται σε πιο στενή επαφή με τους πολίτες. Και εδώ έρχεται και η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συζητήθηκε αυτό το θέμα και στο παρελθόν με την συμμετοχή της Πρόεδρου σας σε μια συνάντηση μαζί με την κυρία Μαγκίνες, την κυρία Γκυγιόμ, τον Αντιπρόεδρο κ. Κατάιν σε σχέση με το συντονισμό για το επενδυτικό σχέδιο. Πώς θα ευδοκιμήσει με κοινέ προσπάθειες, γιατί είναι η πρώτη προτεραιότητα της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου και αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να ανοίξουμε το διάλογο αυτό σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου, να προσκαλέσουμε ε, εκπροσώπους του Κοινοβουλίου στον διάλογο που κάνουμε με τους πολίτες και στις εκδηλώσεις μας ή στην εκκίνηση συγκεκριμένων σχεδίων που εμπλέκουν το Ταμείο Επενδύσεων. Υπάρχει λοιπόν πολύ έφορο έδαφος για συνεργασία. Ελπίζω λοιπόν να θα μπορέσουμε στο υπόλοιπο τμήμα της θητείας μας να το επιτύχουμε αυτό. Αυτός ο διάλογος με τους πολίτες ήταν ουσιαστικός. Είχαμε 50 τέτοιες εκδηλώσεις μέχρι τώρα που παρουσιάστηκαν στις εθνικές τηλεοράσεις. Είχαμε παραδείγματος χάρη αυτό το, την εκδήλωση στην αρχή της έκθεσης του Μιλάνου με την παρουσία της κυρίας Μογκερίν και του κυρίου Σούλτς και θα υπάρξουν και άλλες ε, εκδηλώσεις. Υπήρξαν πολλές εκδηλώσεις όπου τα μέλη του Κοινοβουλίου έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Και θυμόσαστε ότι ο πρώτος Γιούνκερ ήταν παρόν στον διάλογο που έλαβε χώρα στο Μποζά στις Βρυξέλλες πριν από δύο εβδομάδες αμέσως μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι όταν ήταν ε, η, ε, ο συνεργασμό ασφαλείας σε πολύ υψηλό επίπεδο στις Βρυξέλλες και ήρθε σε επαφή με τους πολίτες. Κάτι ακόμα που θέλω να πω γιατί ε, το είδα από τον κύριο Μάλινοφ, είναι η πρωτοβουλία πίσω στο σχολείο. Είναι μια κοινή εμβληματική πρωτοβουλία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 700 μέλη της Κομισιόν ή του Κοινοβουλίου ή άλλοι ε, εθνικοί αξιωματούχοι πηγαίνουν πίσω στα σχολεία τους και συναντήσανε συνολικά 62.000 μαθητές. Και ο κύριος Μάλινοφ έχει συμμετάσχει σε αυτή την ε, ε, πρωτοβουλία. Ξέρω ότι όλοι σας γυρίζετε στα σχολεία σας, στις εκλογικές περιφέρειές σας, αλλά ο σκοπός είναι να το κάνετε αυτό με θεσμικό τρόπο. Επίσης είναι σημαντικά τα πολιτιστικά δρόμενα. Εμείς έχουμε κάποιες πρωτοβουλίε που έχουν σαν τίτλο «Ο Ευρωπαϊκός Δημόσιος Χώρος» και γίνεται στις ε, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τα γραφεία του, της Κομισιόν, μία σειρά από τέτοιες εκδηλώσεις. Αναφέρθηκα στις ε, εθνικές αντιπροσωπείες της Κομισιόν, δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά είναι κέρι εταίροι για το Κοινοβούλιο, επί το οποίο Πάντα είμαστε εδώ στη διάθεσή σας, αλλά και οι εθνικές μας αντιπροσωπείες έχουν αναλάβει το έργο της στενής συνεργασίας με το Κοινοβούλιο και τα Γραφεία Πληροφοριών του Κοινοβουλίου και ένα από τα στοιχεία σε αυτή τη συνεργασία είναι η χρήση των νέων κοινωνικών μέσων διαδικτύωσης όπου έχουμε κοινά σχέδια και νομίζω τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά και μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερα τα πράγματα. Για το σχέδιο επενδύσεων, για τη συνέχιση σε σχέση με το σχέδιο επενδύσεων και τη συνάντηση που είχαμε για την καλύτερη επικοινωνία, προετοιμάσουμε κάτι αντίστοιχο για άλλε προτεραιότητε του χρόνου και είμαστε σε επίπεδο συζητήσεων μαζί σας για τα θέματα τα οποία πρέπει να είναι το κέντρο της επικοινωνίας μας στο μέλλον. Εν τέλει, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτή η πρώτη συζήτηση καταδεικνύει σε μένα τουλάχιστον ότι έχουμε πολλά κοινά στοιχεία. Είναι πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε από κοινού, μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα. Αν εστιάσουμε στον ειδικό ρόλο που έχουμε, δεν χρειάζεται να γίνονται αυτά με τυπικές συμφωνίες και διαδικασίες, μπορούμε να τα κάνουμε με πρακτικό και πραγματιστικό τρόπο συνεργασίες και βασίζομαι ιδιαίτερα στην υποστήριξή σας, ιδίως για να μπορούμε να είμαστε από κοινού ενεργοί σε διάφορε εκδηλώσει στα Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Thank you. Thank you so much. Και εμεί ευχαριστούμε για αυτέ τι επεξηγήσει. Έχω πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις, αλλά θα δώσω πρώτα το λόγο στους συναδέλφους. Η Αντιπρόεδρος Σουιντρόβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η συνεργασία μεταξύ της αντιπροσωπείας του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Κοινοβουλίου λειτουργεί άριστα στην Τσεχική Δημοκρατία. Οργανώνται διάφορες εκδηλώσεις μαζί και εγώ συμμετείχα σε διάφορες εκδηλώσεις, εξακολουθώ να συμμετέχω. Μία από τις ε, δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου θα ξεκινήσει από τον επόμενο χρόνο και θα είναι ένα βραβείο, ε, έχουμε το Lux Film Prize μέχρι τώρα, κοινό βραβείο από του χρόνου, θα πρέπει να αυτό το βραβείο το κινηματογραφικό σαν μια κοινή δραστηριότητα μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωκοινοβουλίου είσαστε ενημέροι επ' αυτού. Και έτσι θα γίνει. Εμείς θα θέλαμε το Ευρωκοινοβούλιο να εξακολουθεί να δραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή να χρησιμοποιείται σαν ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ των βουλευτών και των πολιτών. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Άλλοι συνάδελφοι, ορίστε. Σαμπίν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έλευσή σας ενώπιον της Επιτροπής μας για να μας παρουσιάσετε τις σκέψεις για μια καλύτερη επικοινωνία. Εγώ έχω πάντα την εντύπωση και αυτό το έχουμε συζητήσει εδώ και πολλά χρόνια στην Επιτροπή μας ότι πάρα πολλές από τις πολύ καλές ιδέες που υπάρχουν τελικά δεν φτάνουν τον ευρύ πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αυτό πρέπει να μας ε, απασχολήσει είναι το πώς θα πλησιάσουμε όχι μόνο αυτού, οι οποίοι ήδη γνωρίζουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι εν του τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν περισσότερε πληροφορίε, αλλά να μπορέσουμε να πλησιάσουμε και του άλλου ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν ιδέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην καθημερινή του ζωή, γιατί τα μέσα ενημέρωση δεν λένε τίποτα για τα θέματα αυτά τι περισσότερε φορέ για του πολιτέ. Λοιπόν, να έχουμε μια στρατηγική επικοινωνία για του απλού ανθρώπου για όλους τους πολίτες της Ευρώπης, ακόμα και για αυτούς οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένω ακόμα από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια <clears throat> στρατηγική που θα βελτιώσει τα πράγματα. Καλές είναι οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά δεν πλησιάζουν, δεν φτάνουν όλο τον πληθυσμό. Απλώς ενδιαφέρουν ένα μονάχα τμήμα του πληθυσμού. Εμάς Μα ενδιαφέρει να μπορέσουμε να φέρουμε στον απλό άνθρωπο αυτό που κάνουμε στην Ευρώπη σε καθημερινό επίπεδο. και εγώ σκέφτομαι το τι μπορούμε να κάνουμε και το τι κάνω εγώ στην ε, Γερμανία. Εμείς έχουμε κάνει πολλά πράγματα μέσα από τα σχολεία. Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί δεν υπάρχει μια μεγαλύτερη επαφή των διαφόρων φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα σχολεία, με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θα πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσει πραγματικά το πρόβλημα αυτό να φτάσουμε τους απλούς ανθρώπους, όχι μόνο αυτούς οι οποίοι είναι ήδη ενθουσιασμένους με την Ευρώπη, αλλά αυτούς οι οποίοι δεν έχουν μέχρι στιγμής κανένα κίνητρο να διαφερθούν για την Ευρώπη. Ευχαριστώ Σαμπίν. Υπάρχει άλλος που θέλει να μιλήσει. Ο κ. Κανδοζιεύκη. Παρόμοια ερώτηματα έχω. Όλοι είχαμε την εντύπωση ότι υπάρχει τεράστιο χάσμα μεταξύ των προσπαθειών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, προσπάθεια για πλησίασμα των πολιτών και απ' την άλλη να μην υπάρχει επαρκής γνώσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είναι, πώς λειτουργεί, τι κάνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. In, ε, among... Ε, για τους απλούς πολίτες δεν υπάρχει η γνώση αυτή. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί. Μεγάλο ποσοστό των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σκεπτικιστές όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξέρουμε αυτό. Είδαμε τι έγινε σε εκλογές στη Γαλλία και όχι μόνο. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα και στο Κοινοβούλιο ότι δεν καλούμε ε, προσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων σε συνεδρία των σκιωδών. Είναι καλή λύση αυτή όταν έχουμε τέτοια προβλήματα. Και για τον γενικότερο πληθυσμό ισχύει αυτό. Τους σκεπτικιστές μεταξύ των πολιτών. Τι κάνουμε για αυτούς. Και στην εκλογική μου περιφέρεια υπάρχουν πολλοί σκεπτικιστές και θα θέλω να συναντήσουν κάποιον την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κύριο Γιούνκερ Φερρυπίν. Να του υποβάλουν ερωτήσεις. Τι γίνεται με το LuxLeaks Φερρυπίν. δεν έχουν όμως τη δυνατότητα να μιλήσουν με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι μόνο σε επίσημες εκδηλώσεις, αλλά να ξεκινήσουν πολιτική κουβέντα με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Μαραγάλη έχει το λόγο. Εγώ δεν θα λάβανα το λόγο κυρία Πρόεδρε, αλλά μετά από αυτά που άκουσα στις ε, δύο τελευταίες παρεμβάσεις ένιωσα την ανάγκη να πω και εγώ τα ίδια πράγματα. Να πω ότι ότι βλέπω και εγώ τη σχέση Κομισιόν και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό το πρίσμα της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναρωτιέμαι λοιπόν σε ποιο βαθμό το παιχνίδι συνίσταται στο να μειώνουν τα κράτη-μέλη τη συμμετοχή τους χρηματοδοτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ προσπαθούν να αυξήσουν τα χρήματα τα οποία παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε κρίνουν, κρύβουν τα θετικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξέρουν τα αρνητικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό φυσικά έχει τα αποτελέσματα που γνωρίζουμε και εγώ ξέρω ότι δεν είναι καθόλου εύκολος ο ρόλος σας ως υπεύθυνο επικοινωνίας από την πλευρά της Κομισιόν. Αλλά είναι φανερό ότι υπάρχει μία αντίφαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρνει να εξηγήσει ούτε να παρουσιάσει στους πολίτες το γενικό συμφέρον των Ευρωπαίων. Ο πολίτης δεν καταλαβαίνει καν ότι υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Απλώς έχουμε να κάνουμε ένα αριθμητικό άθροισμα εθνικών συμφερόντων που σχεδόν ποτέ δεν καταφέρουν να πετύχουν κάτι καλύτερο. Πού βρίσκεται λοιπόν το εθνικό, το ευρωπαϊκό συμφέρον σε ό,τι αφορά τον τομέα της φοροαποφυγής των δράσεων των κρατών μελών που δίνουν φορολογικές ελαφρύνσεις μεγάλες επιχειρήσεις. Πού βρίσκεται εδώ η επικοινωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά. Γιατί πολλές φορές προτιμάει να συγκαλύψει τα έσχη τα οποία συμβαίνουν και όχι να υποστηρίξει το γενικό συμφέρον. Και επομένως ένα τμήμα της ε, εξήγησης των αποτελεσμάτων που είχαμε χθες στη Γαλλία βρίσκεται εκεί. Υπάρχουν ε, λόγοι ουσίας, αλλά υπάρχουν και λόγοι που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση την κρίση, την οικονομική και άλλα προβλήματα που οδηγούν σε μεγαλύτερο ευρωσκεπτικισμό. αλλά υπάρχει μια έλλειψη ουσιαστικά εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εαυτό της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει μια πολιτική επικοινωνίας για τον εαυτό της. Άλλο είναι να κάνετε διοργανώσεις, να εξηγείτε συγκεκριμένα προγράμματα. Πρέπει να έχετε μια επικοινωνία για τον εαυτό σας. Ευχαριστώ κύριο Μόργανο και κλείνουμε τις παρεμβάσεις. Eh, και εγώ δεν ήθελα να μιλήσω, αλλά οι συνάδελφοι προέβησαν σε μια εμβάθυνση την οποία συμμερίζομαι. Πολλέ από τις δραστηριότητε που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρύβονται είτε σε έναν κόνο σκιά ε, και δεν είναι γνωστά τα γεγονότα και τελικά πράγματι τα, οι διάφοροι εθνικοί φορεί βασίζονται σε εθνικά στοιχεία και τα προβάλλουν. Υπάρχει διαφορά μεταξύ εκείνων που αποφασίζονται και της επίγνωσης αυτού που αποφασίζεται και πώς γίνεται αποδεκτό. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των δραστηριοτήτων των Εθνικών Κοινοβουλίων σήμερα αντιστοιχεί και σε αυτά που αποφασίζονται εδώ, αντικατοπτρίζει αυτά που αποφασίζουμε εδώ. Έχω μία έκκληση να κάνω. Έχω την εντύπωση ότι αν στα πλαίσια της επικοινωνίας δεν ξεκινήσουμε να επιτρέπουμε στους πολίτες να παρακολουθούν την πορεία των, της νομοθεσίας, τι συζητάμε, σιγά σιγά να βλέπουν την πορεία. Ποια, ποιος είναι ο θετικός αρνητικός αντίκτυπος των αποφάσεών μας. Τι διακυβεύεται, έχω την εντύπωση ότι ο πολίτης θα περιορίζεται στο να ενημερώνεται μόνο για τις αποφάσεις και να μην μπορεί να δώσει περισσότερη προσοχή που απαιτείται η προσοχή ούτως ώστε να λειτουργεί σωστά και το δημοκρατικό σύστημα που είναι και το ίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα. Στατηγική σημασία. Στο πρώτο. Τα καθήκοντα. Αρμοδιότητα της επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απορρέει από το ότι είναι θεματοφύλακα των συνθήκων και της ταυτότητας. θέλει να δώσει ορατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει επίσης να εξακριβώνει ποια εικόνα προβάλλεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εκεί εξαρτώνται και τα μέσα που τα χρησιμοποιούνται και εικόνα αυτά προβάλλεται. Είναι πολύ σημαντικό. Ποιε προτεραιότητε καθορίζονται πέρα από το περιεχόμενο των προγραμμάτων. Σαφή τα προγράμματα είναι οι προτεραιότητε του Juncker. Οι βασικοί προτεραιότητες. οι βασικέ προτεραιότητε αλλά πρέπει να πούμε σε βάθος. σε Συζητάμε λοιπόν την ίδια την ταυτότητα της Ένωσης, τη χρησιμότητά της, την αναγκαιότητα ύπαρξής της. Υπάρχει κάποια αντίφαση. Από τη μία πλευρά 75% των νόμων των κρατών μελών απορρέουν ευρωπαϊκές οδηγίες και από την άλλη λένε ότι δεν μετράει τίποτα η Ευρώπη. Και υπάρχει και άλλο μεγάλο θέμα της αποστασιοποίησης και της απογοήτευσης όσον αφορά την Ευρώπη. Το βλέπουμε και στα πολιτικά αποτελέσματα τα πρόσφατα. Ερώτηση. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται πολύ στην επικοινωνία. Σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί στο μέλλον, τι εκστρατεία θα ακολουθήσει, υπάρχουν στόχοι εκστρατεία για τις νέες γενιές. Ποιους target έχει θέσει. Κάποτε γινόταν εκστρατείες όσον αφορά το κόστος της μη Ευρώπης. Όταν αφισβητείται η Ευρώπη πρέπει να υποθεί με σαφήνεια πόσες περισσότερες δυσκολίες θα είχαμε αν δεν υπήρχε περισσότερη Ευρώπη. Τρίτον, οι πόροι για την επικοινωνία. Υπάρχουν λεπτομέρειες όσον αφορά τη DGCOM, τι έγινε κατά το παρελθόν ή δεν υπάρχουν. Για τη συμμετοχή των βουλευτών σίγουρα βελτιώθηκε σε εθνικό επίπεδο. Υπενθυμίζω ότι μέχρι πριν από μερικού μήνε, όταν οι επίτροποι συναντιόνταν με του ε, πολίτε διαφόρων χωρών μελών, καλούνται οι κυβερνήσει, αλλά όχι οι ευρωβουλευτέ, οι, συγγνώμη, οι εθνικοί βουλευτέ. Νομίζω ότι αλλάζει. Και στη συνάντηση που θέλαμε να κάνουμε μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη DGCOM, με το Ευρωκοινοβούλιο και με την Προεδρία και τι Επιτροπέ, κινούμεθα προ τα εκεί να υπάρχει συμμετοχή των βουλευτών. Είναι σημαντικό αυτό στο μέλλον να γίνει. Να δούμε ποια είναι τα ισχυρά και τα στενή σημεία της προσπαθίας που καταβάλλετε. Ποια μέσα έχουμε στη διάθεσή μας. Είπατε ότι η Connect ασχολείται με το Euronet και το Euronews. Τι εργαλεία έχει η Digicom όταν η Connect έχει πάρει τα εργαλεία. Έχετε διασύνδεση με την άλλη γενική διεύθυνση είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων αυτές οι ερωτήσεις που θέτω. Thank you very much, President. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα προσπαθήσω να σας απαντήσω όσο μπορώ καλύτερα. Πρώτον, την κυρία Σόλη Ρόβα για το βραβείο Λούξ. Ξέρω ότι η χειρότερη δυνατή απάντηση που μπορεί να δώσει ένας γραφειοκράτης είναι δεν είναι δική μου δουλειά αλλά κάποιο άλλο. Δυστυχώς όμως σε αυτή την περίπτωση ισχύει. Ξέρω βέβαια, έχω ακούσει για αυτό το βραβείο και θα αναφέρω στους σχετικούς συναδέλφους μου. Αλλά δεν έχω την δικαιοδοσία να σας απαντήσω ή να αποφασίσω γι' αυτό. και στη Γενική Διεύθυνση Connect έχουμε καλή συνεργασία. Και για Μπεχάιαν τώρα. Βασικό το ερώτημά σας. Εγώ σας έδωσα μια σύντομη δεκάλεπτη περιγραφή Έχουμε και επιτόπου υπεύθυνους πληροφόρησης δεν είναι υπάλληλοι της Κομισιόν αλλά πληρώνονται από κάποια στοιχεία του προϋπολογισμού και τους ενθαρρύνουμε να συνομιλούν με τους πολίτες καθημερινά με τους απλούς πολίτες. Είναι καμιά 700 αριά και το σύστημα αυτό δουλεύει πάρα πολύ καλά όσο για τους συναδέλφους στην Επιτροπή των Περιφερειών και αυτοί παίζουν σημαντικό ρόλο. Και αυτοί. Ότι δεν περνάει το μήνυμα, ναι, και εγώ το βλέπω πολλές φορές. Μόλις γίνει μία πρόταση, σε λίγο το κοινοβούλιο να συζητάει την εγκρίνη το Συμβούλιο, αλλά καμιά φορά η δυσκολία είναι ότι οι πολίτες Συγχίζονται, συγχέονται, μπερδεύονται. Μπορεί να κάνει ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος κάποια συνέντευξη τύπου, αλλά μετά θέλει το κοινοβούλιο να αλλάξει τη θέση. Υπάρχει και αυτό το διαθεσμικό δηλαδή επικοινωνιακό πρόβλημα που μπερδεύει τους πολίτες. Αυτό είδα εγώ, αυτό είδα, αυτό είδα, αυτό είδα και στην προηγούμενη θέση μου. Αν τον κύριο Κρανοντεύσκη για τους ευρωσκεπτικιστάς. Εμείς δεν τους φοβόμαστε. Θέλουμε να συζητήσουμε και μαζί τους εφόσον θέλουν να μας ακούσουν με βάση γεγονότα για τις προτεραιότητες μας και τα προγράμματά μας. Ο κόσμος δεν είναι ασπρόμαυρο το ξέρουν αυτό οι πολίτες. Και είναι μεγάλη πρόκληση για όλους μας και για την Καμισιόν και για το Κενοβούλιο. Αλλά υπάρχουν και τα κράτη-μέλη. Αυτά που αποφασίζουν τα τρία όργανα πρέπει να συναποφασιστούν και από τους, τις δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις και κοινοβούλια των χωρών μελών. Δεν είναι σωστό να λένε αυτό που λένε συχνά. Εμείς θέλαμε κάτι διαφορετικό αλλά έτσι αποφάσισαν οι Βρυξέλλε. Ναι, Για ε, τον κύριο Μαραγκάου για τη φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή. Όχι, δεν αποφεύγουμε το θέμα. Αποφεύγουμε. Πολύ σύντομα καταλή... ε, προτείναμε μία δέσμη φορολογική και γι' αυτό δεν συμφωνώ μαζί σας αλλά συμφωνώ ότι υπάρχουν προγράμματα που χρειάζονται πρόσθετη προσπάθεια επεξήγησης από τους, προς τους πολίτες και αυτά που είπε ο κύριος Μοργκάνο καμιά φορά η διατύπωση που χρησιμοποιούμε είναι πρόβλημα να μην κρυβόμαστε εδώ γράφουμε προτάσεις σε σπασμένα αγγλικά ή γαλλικά και μεταφράζονται μετά στις εθνικές γλώσσες και καμιά φορά χρησιμοποιούμε τεχνική γλώσσα ή ακρονίμια ακόμη και οι δημοσιογράφοι ακόμη και οι μόνιμοι ανταποκριτές δεν καταλαβαίνουν οι πολιτικοί πρέπει να μιλάνε αλλιώς τα μέσα ενημέρωσης από ό,τι μεταξύ τους. Να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών, τη γλώσσα του λαού. Το μήνυμα λοιπόν δεν μεταφέρεται άμα δεν υπάρχει και η σωστή γλώσσα, ούτε τα αισθήματα. Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στις προσπάθειες για τους νέους. Οι έχουν αυτή την πρωτοβουλία επιστροφή στο σχολείο, τη στήριξη των διδασκάλων, ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών, επισκέψεις επιτρόπων σε πανεπιστήμια. Ξέρουμε ότι δεν αρκούν όλα αυτά με ναι, λοιπόν. ναι, υπάρχουν και τα κοινωνικά μέσα, ναι. Και για το roaming, από το roaming είχαμε μεγάλη επιτυχία, κάτι πολύ συγκεκριμένο και που ήθελαν οι πολίτες και ιδιαίτερα οι νέοι. Το θεωρούν κάτι συγκεκριμένο που μπορεί να κάνει η Ένωση. Πολύ ωραία πέρασε αυτό. Για τον προϋπολογισμό χάσαμε μόνο δύο προγράμματα αλλά δεν έγιναν γενικά περικοπές. Για του χρόνου χάρη στη στήριξή σας αυξήθηκε ο προορισμός μας κατά 6% και υπάρχει και ο ειδικό προϋπολογισμός για την corporate communication για να καλυφθεί η επικοινωνία για τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Εκεί μπορούμε να πετύχουμε μια συνέργεια που, με την οποία θα συμφωνούσαν και ο κύριος Μοργκάνο και άλλοι. Αλλά τα λεφτά δεν λύνουν αυτά τα προβλήματα. Μπορεί να βοηθήσουν, αλλά χρειάζεται πολιτική θέληση. Ξέρω ότι και εμείς και εσείς την έχουμε και την έχετε, άρα όλα πάνε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Υπολογίζουμε στην υποστήριξή σας και στο μέλλον για τη γενική σας διεύθυνση, μεταξύ γενικής σας διεύθυνσης και κενοβουλίου. Ευχαριστούμε πολύ και γκράτζι μίλε. Τώρα λοιπόν με τους συναδέλφους της Επιτροπής Πρέπει να πω το εξή. η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου από τις 3 μέχρι τι 6.30 το απόγευμα. Ε, πόσο είναι η τελευταία συνεδρίαση πριν από τα Χριστούγεννα. Θέλω να σε απευθύνω πολλές ευχές σε εσάς, στις οικογένειές σας, στους συναδέλφους βεβαίως, σε όλους τους policy advisors, βοηθούς, γραμματεία και βέβαια σε όλους που είστε εδώ παρόντες. Πάρα πολλές καλές ευχές Δουλέψαμε πολύ αυτό το χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια. Πιστεύω ότι συμβάλαμε κατά σημαντικό τρόπο με τα θέματα που εξετάσαμε και πιστεύω ότι σήμερα κλείνουμε το χρόνο με μεγαλύτερη γενική επίγνωση ότι χρειάζεται επένδυση στον πολιτισμό και στην παιδεία. Είναι αναγκαίο. Όχι μόνο για τα θέματα που μας αφορούν, αλλά επειδή χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα για τις νέες γενιές. Έχουμε μπροστά μα ένα χρόνο με πολλή δουλειά. Ευχαριστώ όλου. Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο ο καινούριο χρόνο. Θα παρακαλούσα τώρα του συντονιστέ να παραμείνουν στην αίθουσα. Θα ξεκινήσουμε αμέσω τη συνεδρίαση των συντονιστών. Όποιο πρέπει να αποχωρήσει, το κάνει τώρα παρακαλώ. Σα αποχωρήσει από την αίθουσα για να ξεκινήσουμε αμέσω τη συνεδρίαση των συντονιστών. Έχουμε καθυστερήσει, βλέπετε. Επτά λεπτά. Όχι τόσο πολύ, τόσο πάνω. Έχουμε καθυστερήσει λίγο. How many? Three? Three. Uh, three. We uh, three, four and five. Okay. Five coordinators and uh,